willkommen zur Sitzung heute Nachmittag. Und es ist mir eine besondere Freude, den Kommissar... Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε την απευθυνή μας συνεδρίαση και με μεγάλη χαρά καλωσορίζω σήμερα τον Γιάννη Ποτόσκι για την ανταλλαγή απόψεων Θέλουμε με τον κύριο Επίτροπο ναι. να έχουμε έναν τακτικό διάλογο και βεβαίως μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να, ακούσουμε στην αρχή του χρόνου τι μας περιμένει και το πρόγραμμα των επόμενων έξι μηνών. Είχαμε προτείνει να οργανώσουμε τη συζήτηση κάπως για να μπορέσουμε και να εμβαθύνουμε στα διάφορα θέματα Τρία είναι λοιπόν τα κύρια θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Καταρχάς οι, αποτελεσ... οι... οι πόροι. Δεύτερον, προτεραιότητες και τρίτον, εφαρμογή, υλοποίηση και τέταρτον, διάφορα, όλα τα υπόλοιπα θέματα. Η γραμματεία έχει λοιπόν συντάξει έναν κατάλογο μιλητών 27 ερωτήσεις. Προς το παρόν έχουν εγγραφεί. Ο κύριος Ποτότσνικ πρέπει ακριβώς στις 4.30 να φύγει. Ένα λεπτό με ενάμιση έχει ο κάθε, το κάθε μέλος, ο κάθε συνάδελφος να θέσει ερώτημα. Δεν θέλω λοιπόν να σας ε, καθυστερήσω, παρακολουθήσαμε και τις συνεδρίες των αντιπροέδρων και είδαμε ότι ε, είχατε το ρόλο του συντονιστή, του facilitator. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση και η συνάδελφός μας, η κυρία Χέντεγκερ, είχε επίσης μια επιτυχή συμμετοχή στο Κανκούν και η πολυμερής αυτή η διαδικασία, όλες αυτές οι διαβουλεύσεις ε, προχώρησαν το 2010. Και γι' αυτό δίνω απευθεία το λόγο στον κύριο Επίτροπο και αρχίζω με τον πρώτο γύρο. Ε, οι πόροι, πόροι, επαρκείς πόροι, επάρκεια πόρων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Short remark, uh, let's say horizontally on the issues from the environmental side and immediately then I will switch to the resource efficiency, which is our first topic.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 The Commission will adopt tomorrow a communication on the resource efficiency flagship, which will set the scene for all the different initiatives to be adopted in 2011 and 2012 within this framework. This communication will show that... Αυτό θα δείξει ότι η αποτελεσματικότητα των πόρων δεν είναι μόνο θέμα της Κομισιόν, αλλά και πολιτική ολόκληρη της Ένωσης θα επιτρέψει την καλύτερη συμπερίληψη των συμπεριβαλλοντολικών στόχων σε άλλα προγράμματα μεταξύ των οποίων και την οικονομική ανάπτυξη. Μόλις ένα χρόνο πριν δεν αναφερόταν καν η έννοια αυτή της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων. Ελπίζω να μπορέσει να συνεχίσει να συζητιέται, πράγμα που δεν ήταν καθόλου σίγουρο. Πρέπει βέβαια για να γίνει πράξη να γίνουν ακόμη πολλά. Θα ήθελα μαζί να τα κάνουμε όλα αυτά γιατί χρειάζεται συνδυασμός προγραμμάτων για να τροποποιηθεί ολόκληρη η οικονομία μας να μεταμορφωθεί και γι' αυτό χρειάζεται η πλήρη στήριξη της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου. Εγώ με τις υπηρεσίες μου επεξεργάζομαι έναν οδικό χάρτη για μια πιο αποτελεσματική χρήση των ε, ενεργειακών πόρων στην Ευρώπη. Θα αποτελέσει αυτό ένα πρόσθετο εργαλείο για, τις αναπτυξια, για τα αναπτυξιακά προγράμματα. Δηλαδή θα αναφέρει και λεπτομερείς προτάσεις. Εμείς στην Κομισιόν αλλά γενικότερα στην Ευρώπη έχουμε κάνει μεγάλες πρόοδους του τελευταίους 12 μήνες στις συζητήσεις μας για την αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων. Και είπαμε ότι η καλύτερη διαχείρισή τους είναι ουσιώδης παράγων για το μέλλον του πλανήτη. Συμφωνήσαμε ότι μια οικονομία με καλύτερη χρήση των πόρων είναι βασικός τρόπος για να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και επίσης συμφωνήσαμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε αποτελεσματικά για συνδυασμό προγραμμάτων και εθνικά ώστε να επιτευχθούν οι αλλαγές που χρειάζονται. Τώρα όμως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα που θα αποφασίσουμε θα ανταποκρίνονται και στους στόχους μας. Να μην υποτιμήσουμε το, την κλίμακα των αλλαγών που χρειάζονται, αλλά να χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον τέσσερις μεθόδους για την μετατροπή της ευρωπαϊκής οικονομίας σε πιο αποτελεσματική. Πρώτον, να εφαρμοστεί η νομοθεσία που έχουμε ήδη υπογράψει για τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση. Αυτό θα σήμαινε ότι θα βελτιώναμε πολύ τη χρήση των πόρων και θα ε, βελτιωνόταν και η κατάσταση της απασχόλησης. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να υπάρξει πλήρης εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη τα τελευταία πέντε χρόνια. Και αυτό θα παραμείνει προτεραιότητα και τον επόμενο χρόνο για μένα και για την Επιτροπή ολόκληρη και επομένως η εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα καθώς και η πρόσφατη αναθεώρηση άλλων οδηγιών θα α, μπορέσουν να αποτελέσουν σημαντικά βήματα πρόοδου. Περισσότερα βέβαια πρέπει να γίνουν και για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και για τη μείωση των χωματερών. Η λύση, είμαι πεπισμένος, δεν έγκυται μόνο στην νομοθεσία αλλά και στη δημιουργία νέων αγορών για δεύτερη χρήση των υλικών για να υπάρξουν έτσι λιγότερα απόβλητα. Δεύτερον, πρέπει η αγορά να οδηγηθεί με εργαλεία που να είναι ακριβώς της αγοράς, παραδείγματο χάρη τιμές που να ανταποκρίνονται περισσότερο στο πραγματικό κόστος και η φορολόγηση να μετατοπιστεί για να δοθεί ένα κίνητρο οι οικονομίας μας να κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε βέβαια να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλου είδους φορολόγηση. Συζητώντας με τον συνάδελφό μου σε μέταν πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό καλύτερα είδαμε ότι πρέπει σύντομα να αρχίσουμε να εργαζόμαστε για την κατάργηση των βλαβερών επιχορηγήσεων. Φέτος θα γίνει η πρώτη μελέτη μας για αυτό το λεγόμενο Smart Fiscal Consolidation πρόγραμμα. Τρίτον, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα εργαλεία που ήδη έχουμε αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε καλά ή απαρκώς. Οι οικοετικέτε και άλλα τέτοια προγράμματα οι εργαλεία μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική αλλαγή και για τις επιχειρήσεις και για τα κράτη. Παράδειγμα, θέτοντας κριτήρια οικολογικής αποτελεσματικότητας μπορούν μερικά προϊόντα να γίνουν πιο αποτελεσματικά, να μειωθεί η εκπομπή αερίων και μέχρι το 2020 να υπάρξουν εξοικονομήσεις ανά χρόνο σχεδόν 13% της τωρινής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Βέβαια τέτοια εργαλεία βιώσιμης παραγωγής είχαν ήδη ακουστεί από το 2008 αλλά πρέπει να επεκταθούν όπως με το να περιλαμβάνουν οι σχετικές οδηγίες νέες ρήτρε. Όλοι αρχίσαμε μαζί να σκεφτόμαστε 2012. τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος SEP για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμη περισσότερα αποτελέσματα φέτος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά θα είναι βασικός παράγοντας στη διαβούλευση αυτή. Και τέλος, τέταρτο δηλαδή μάλλον, πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη προσέγγιση για την επίτευξη βιώσιμων μεθόδων διαχείρισης και αποτελεσματικότητας. Πέρα και από την καθαρή περιβαλλοντολογική πολιτική. Αυτό θα απαιτούσε μια μεγαλύτερη, ένα, μια μεγαλύτερη παιδαγωγική προσπάθεια, πράγμα που είναι δύσκολο εφόσον οι περισσότεροι προσέχουν μόνο τα δημοσιονομικά αυστηρά. Αλλά η διαδικασία του 2020 πρέπει να μας δώσει μια ευκαιρία να τα καταλάβουμε όλα περισσότερο. Η αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων που διαθέτουμε μέσα στην οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης αλλά και μέσω συγκεκριμένων εργαλείων πολιτικής είναι μια καλή ευκαιρία παραδείγματος χάρη. Οι δημόσιες... Ε, Here I also προμήθειες θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν και θα το τονίσω και στους συναδέλφους μου καθώς και σε εσάς ότι πρέπει να δούμε ακριβώς ποια είναι η αποτελεσματικότητα της δουλειάς μας και όλο της κάθε επιτροπής και γενικής διεύθυνσης. Το πρώτο έτος λοιπόν της εντολής μου μου δίδαξε ότι ανοίγει μία νέα εποχή για το περιβάλλον. Από πολιτική κατακαιρματισμένοι πρέπει να οδηγηθούμε σε μια πιο συστημική πολιτική που να ανταποκρίνεται στο πολύπλοκο χαρακτήρα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το περιβάλλον και η κοινωνία μας. Και γι' αυτό πρέπει να εντατικοποιήσω την εργασία μου μαζί με άλλους επιτρόπους. Παραδείγματος χάρη είχαμε πολύ ενθαρρυντική συζήτηση την περασμένη εβδομάδα για την ποιότητα του αέρα με στόχο να αυξηθεί η συνειδητοποίηση του προβλήματος και να δούμε πώς θα μπορούσαμε συνδυασμένα να κάνουμε κάτι. Πρέπει τα προγράμματα να συνδυάζονται για τέτοια προβλήματα. Η μετατροπή της οικονομίας σε βιώσιμη ανάπτυξη είναι κάτι που πρέπει να το αρχίσουμε από τώρα ώστε μέχρι το 2020 να έχουμε προχωρήσει προς την κατεύθυνση που θέλουμε για την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο. Δύσκολο έργο βέβαια, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα αν μπορώ να υπολογίζω στην υποστήριξή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επίτροπε κύριε Κοτότσνικ. Βεβαίως η Επιτροπή μας είναι πρόθυμη να υποστηρίξει αυτή την πολιτική μέσα στο πλαίσιο της οικολογικής πολιτικής προστασίας περιβάλλοντος και βιοπικιλότητας. Προχωρούμε συστηματικά ε, και ανακλάδω στην πολιτική αυτή ε, για να εξασφαλίσουμε την σωστή απόδοση, σωστή ε, αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των πόρων το θέμα είναι όχι μόνο η προμήθεια πρώτων υλών, αλλά και η σωστή τους ε, χρησιμοποίηση, ε, το βέλτιστο τρόπο, η βέλτιστη απόδοση αυτών των πρώτων υλών. Δεν θέλω ε, λοιπόν να μακρηγορήσω για να μπορέσω να σας δώσω χρόνο ομιλίας. 1,3 λεπτά έχετε. Ο Ρίχαρτ ένα 1,3. Αυτό είναι το ορισμό κλειδί. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, παρακαλώ διακόψτε με αν ξεπεράσω το χρόνο. Λέει ο κύριος Ζίμπερ, κύριε Επίτροπε, είσαστε συνέχεια βραχνός όταν σας ακούω, άρα λοιπόν αυτό ίσως οφείλεται στην επικοινωνία σας επειδή μιλάτε πολύ. Λοιπόν, ε, θα ήθελα να ξέρω τι θα κάνετε ως Επίτροπος ε, για να ενημερώσετε τους πολίτες όσον αφορά την ε, επάρκεια και σωστή χρήση των ενεργειακών πόρων δεν νομίζω να έχουμε μεταφέρει στον πολίτη αυτά τα οποία επισημούμε να εφαρμόσουμε. Τι θα κάνετε λοιπόν για να ε, φτάσει το μήνυμα και να γίνει κατανοητό από τους πολίτες. Αν δεν καταλάβουν δεν μπορούν να μας υποστηρίξουν. Ειδικά τώρα για την αποδοτικότητα των πόρων ε, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην Ευρώπη. Ε, υπάρχει αυτή η μόνιμη κρίση των ε, εκπομπών ε, και των απορριμμάτων και υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν καν εγκαταστάσεις καύσεως αλλά υπάρχουν πάλι άλλες χώρες οι οποίες ανακυκλώνουν τα απορρίμματα πολύ επιτυχημένα πολύ λοιπόν μεγάλες διαφορές όσον αφορά την ανακύκλωση και χρήση των απορριμμάτων. Ο Μάριο. Ευχαριστώ Επίτροπε. Διάβασα με ενδιαφέρον την τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατηγική ε, σχετικά με την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Από την ανακοίνωση αυτή φαίνεται ότι η ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων δεν έχει ε, προς το παρόν τουλάχιστον ολοκληρωθεί. Υπάρχουν επίσης προβλήματα και σε σχέση με την μετατροπή τους σε ποιοτικό κόμποστ και φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά και σε μία αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την υλή η οποία προέρχεται από την επεξεργασία αυτών των αποβλήτων. Γιατί να μην ξεκινήσουμε με μια νέα οδηγία σχετικά με την υποχρεωτικά επιλεκτική συλλογή των απορριμμάτων, ένα κοινοτικό πλαίσιο συνολικό συνεκτικό που παρέχει σε όλους τους χρήστες του τομέα και στις δημόσιες αρχές τις απαραίτητες εγγυήσεις και προς τους πολίτες ε, ε, σχετικά με την περιβαλλοντική ασφάλεια. Εποφελούμε τις ευκαιρίες αυτής να ζητήσω κύριε Επίτροπε και τις δικές σας ε, εκτιμήσεις σχετικά με το πρόγραμμα που έθεσαν σε εφαρμογή οι αρχές της καμπανίας για να ξεφύγουμε πλέον από το πρόβλημα των απορριμμάτων. Διακόπτη τον ομιλητή ο Πρόεδρος. Ξεπεράσατε το 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ τον κύριο Ποτόσνικ για τον πρώτο του έτος και για τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει ε, ο κύριος Γκερμπράντι. Έχω ορισμένε ερωτήσεις όσον αφορά την αποδοτικότητα πόρων. Υποστηρίζω την κατεύθυνσή σας απόλυτα, αλλά βλέπω και μια άλλη επιλογή, την εξασφάλιση της εισρωής πόρων αυτή τη στιγμή η κατάσταση που έχουμε δεν είναι ικανοποιητική. Θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο αποδοτικοί. Πώς θα μπορέσετε λοιπόν να ε, εμποδίσετε την μετατόπιση από την εξασφάλιση στην σωστή απόδοση, σωστή αποδοτικότητα των πόρων. Ε, όχι μόνο λοιπόν εξασφάλιση αλλά και βέλτιστη αποδοτικότητα. Ε, η κατεύθυνση που ακολουθείτε επικεντρώνεται στις ενεργειακές πηγές και στο νερό, στο, στους υδάτινους πόρους. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να διευρύνετε τους, ε, τα θέματά σας. Και επίσης πώς θα αναπτυχθούν οι περιβαλλοντικοί λογαριασμοί. πιστεύω Πιστεύετε ότι τα, τα μέσα που προβλέπουν για το Life Plus, το Life Sin μπορούν να εφαρμοστούν σωστά από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος, λέει ο κύριος Σάικοτ. Ε, σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε και ειδικά για την κατευθυντήρια γραμμή που θα ανακοινωθεί αύριο για τις νομοθετικές σας προτεραιότητες. Αυτές οι προτεραιότητες θα καλύπτουν όλες τις γενικές διευθύνσεις. Πράγματι χρειαζόμαστε μία κατεύθυνση γενική, μία ομπρέλα αν θέλετε, η οποία θα καλύπτει όλες τις πολιτικές όλα, όλα, όλα αυτά τα, οι ανακοινώσει για την ενέργεια, για την χρήση της γης, ε, για τους υδάτινους πόρους πρέπει να είναι ε, ε συνεπείς ε, με τις κατευθυντήριες γραμμές. Ένας καθαρο, ξεκάθαρος στόχος είναι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε καλύτερα, και να καλύτερα τη, τη γη, έτσι ώστε να συμβαδίζουν οι αποφάσεις με την μεταρρύθμιση της αγροτικής πολιτικής. Ο δικός χάρτης που θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο μπορεί να τα συντονίζει όλα αυτά. Αλλά πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι υπάρχει συνοχή και συνέπεια ε, στην ατζέντα σας, η οποία καλύπτει όλους τους πόρους. Λοιπόν, συνέπεια και συνοχή. Ευχαριστώ. Το ερώτημά, μου, το ερώτημά μου λέει η κυρία Γκέρλινγκ ε, είναι, αφορά την ε, περιβαλλοντική νομοθεσία η οποία είναι, ε, έχει κόστος σοβαρό. Πώς λοιπόν θα εξασφαλίσουμε το, τη ζωή μας σε ένα καλύτερο περιβάλλον, ποιοτικά δηλαδή. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε όλοι ότι αντιμετωπίζουμε μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι γίνεται αυτή τη στιγμή ένας δημοσιονομικός ε, συγκερασμός, ε, μια, ε, ένας περιορισμός γενικά δηλαδή στο, στα δημοσιονομικά θέματα και όμως έχουμε πολλά εκκρεμή ζητήματα στην περιβαλλοντική νομοθεσία όπως τα απόβλητα, στα απορρίμματα, όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και προσπαθούμε να βρούμε πιο έξυπνους τρόπους να χειριστούμε αυτά τα θέματα με λιγότερες δαπάνες, αλλά τότε σκοντάφτουμε σε άλλους ε, κανονισμούς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, π.χ. στον ανταγωνισμό, τους, τους οποίους πρέπει να σεβαστούμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, ζητήσω να, να έχετε πάντοτε υπόψη σας τα οικονομικά θέματα και τα περιβαλλοντικά. Ευχαριστώ. Επόμενος. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Ρόσπαχ. Μόλις αλλάξαμε θέση. Θα ξεκινήσω με κάποιες ερωτήσεις προς τον κύριο Ποτόσνη. Πώς βλέπετε, κύριε Επίτροπε, τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρήπανσης. Δύσκολο. Ιδιαίτερα με τα πλαστικά απόβλητα τα οποία ρίπτονται στη θάλασσα. Πρέπει να υπάρξει μήπως ένα πρόγραμμα δράσης ειδικά για τα πλαστικά που έχουν απορριφθεί στη θάλασσα. Δεύτερη ερώτηση. Για την πολιτική την οποία ακολουθεί η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας σχετικά με τους σπάνιους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιείται από την Κίνα σαν πολιτικό μέσο θα έλεγα. Και τρίτη ερώτηση. Θα υπάρξει ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των φυσικών πόρων. Πιστεύετε ότι υπάρχει επαρκής επαναχρησιμοποίηση τουλάχιστον σε επίπεδο οργανικών αποβλήτων. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ είμαι βραχνή λέει η κυρία Χίμπνερ. Και ε, θα μιλήσει συνάδελφός μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει η κυρία Βίλμοτ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το, το όραμά σας, για το πού θα κατευθυνθείτε. Μιλήσατε για την ε, έγκριση του σημερινού πλαισίου, ε, βεβαίως, ε, αυτό είναι προϋπόθεση. Εμείς θέτουμε τους κανόνες, αλλά πρέπει και να εφαρμοστούν, να υλοποιηθούν και να επιβιώσουν. Ε, ποιες, ποια είναι λοιπόν τα μέτρα τα οποία θα πάρετε, ε, το σκεπτικό δηλαδή που θα ακολουθήσετε Ήδη με άλλους συναδέλφους ε, σας έχω παρουσιάσει την ιδέα μίας κοινωνίας όπου δεν έχουμε όλοι την ανάγκη να αγοράσουμε ηλεκτρικές συσκευές αλλά μπορούμε να τις ε, μισθώσουμε με χρονομερισματική μίσθωση ε, έτσι ώστε να μπορούν και να ανακυκλωθούν με leasing δηλαδή έτσι ώστε θα υπάρχει κοινή ευθύνη του καταναλωτή και του παραγωγού. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει να προχωρήσει μια τέτοια ιδέα. Η Κατρίν Σουλιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι πρώτες ύλε και η ανακύκλωση των αποβλήτων είναι σχετικά θέματα. Ιδιαίτερα θα ήθελα να μιλήσω για τα πλαστικά απόβλητα έχουν διπλό όφελος για ανακύκλωση και ενεργειακό όφελος. Μου φαίνεται σημαντικό να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα απόβλητά μας, αυτά που παράγονται στο έδαφος μας δηλαδή. Ερωτώ λοιπόν, η Κομισιόν έχει καμιά ιδέα για το επίπεδο στο οποίο επιτεύχθηκαν οι στόχοι της συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων και ποια πρέπει να είναι η μελλοντική πολιτική για τη βελτιστοποίηση της ανακύκλωσης αυτής. Όσο για το θέμα των εισαγωγών, μονόπλευρων εισαγωγών από την Κίνα, τι μπορεί να γίνει. Ευχαριστούμε η Μαρίτα Χόιφνερτ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί συζητάμε εδώ για το θέμα της αποτελεσματικότερης χρήσης των πόρων. Ιδιαίτερα δε για τις πρώτες ύλες. Ο Επίτροπος μας ανέφερε έναν κατάλογο όσων πρέπει να γίνουν, καλύτερη χρήση των υπαρχόντων φορολογικών εργαλείων, ανακύκλωση και λοιπά, προμήθειες και δημόσιες προμήθειες και τέτοια. Όλα αυτά πολύ καλά. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι τι πρέπει να κάνουμε, αλλά πώς. Διότι εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο Υπουργών λαμβάνονται αποφάσεις, ε, εγκρίνονται επιχορηγήσεις στα ορυχεία, στα ανθρακορυχεία και αλλού και ξέρουμε πώς λειτουργούν οι αγορές. Είδαμε ποια ήταν η απάντηση της Ρωσίας ως προς την εκμετάλλευση της Αρκτικής. Υπάρχει μια νέα πικιακή θα έλεγα δύναμη η Κίνα και όλα αυτά τα μέτρα αντιφάσκουν με όσα λέμε εδώ. Διότι υπάρχουν πτυχές που, προβλήματος που αφορούν την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό, η Κομισιόν τι πρόκειται να κάνει. Μάλιστα αυτός ήταν ο πρώτος γύρος. Δεν θα είναι ο τελευταίος, θα ξαναμιλήσουμε για αυτά τα ίδια θέματα αλλά ορίστε οι απαντήσεις. Θα αρχίσω με το ερώτημα της, του τρόπου εφαρμογής και των διαφορών που υπάρχουν στην Ευρώπη, στην ε, υλοποίηση και χρήση των πόρων. Έχετε δίκιο στο έκθεση που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα για τα απορρίμματα ε, γενικά αυτό αποδεικνύεται ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ή περισσότερη ενημέρωση των πολι... μέσω των πολιτών με σεμινάρια, επιμορφωτικά, ενημερωτικά ε, και φυλάδια, οδηγίες αλλά και Ε, ενημέρωση ειδικά για τις χώρες που δεν έχουν καταλάβει τι μπορούν να κάνουν. Πέντε. Πέντε χώρες στην Ευρώπη όπου οι χωματερές είναι λιγότερο από 5% και άλλες χώρες στην Ευρώπη οι χωματερές είναι πάνω από 80%. Βλέπετε λοιπόν τις τεράστιες διαφορές. Και από αυτή την έκθεση προκύπτει ότι εάν αυτές οι χώρες πραγματικά αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτά που προτείνει η έκθεση, θα αλλάξει η νοοτροπία, θα αλλάξει ο τρόπος σκέψης και θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν πολύ περισσότερο και καλύτερα τους πόρους. Αλλά χρειάζεται πολύ δουλειά πριν αλλάξει η νοοτροπία, πριν αλλάξει ο τρόπος ε, σκέψης τουλάχιστον στα απορρίμματα ε, και στην ε, ε, χρήση και ανακύκλωση, καύση κλπ. Κάτι προχωράει στην Ευρώπη, κάτι γίνεται. Τώρα, όσον αφορά την, τα βιοαπορρίμματα, ξέρετε το Μάιο το 2010 υιοθετήθηκε μία απόφαση που λέει ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης αυτού του τομέα και, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να βελτιωθεί η οδηγία για τις χωματερές. Ε, ξέρουμε ότι η γνώμη του Κοινοβουλίου διέφερε από αυτήν της, του Συμβουλίου. απευθυνθήκαμε στην Κομισιόν και πολλές φορές εγώ είπα ότι προτείνουμε να καθορίσουμε τα κριτήρια για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ε, κομπόστας για να χρησιμοποιηθούν μίνιμουμ πρότυπα για τη χρήση βιοαπορριμμάτων και για την βελτίωση των ε, συστημάτων αποκομιδής και συλλογής ε, των απορριμμάτων. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία επεξεργαζόμαστε και μελετάμε. Εν εξελίξει λοιπόν. Τώρα, καμπάνια τι Είναι μια μεγάλη ιστορία και δεν υπάρχει γρήγορη λύση με το θέμα της καμπάνια. Είναι δύσκολο το θέμα και ε, συνεχώς ε, είμαστε σε επαφή με περιφερειακές αρχές και πριν από μερικές χώρες ε, λάβαμε, μας ενημέρωσαν για, για, για το νέο διαχειριστικό συμβούλιο πρέπει να δημιουργηθεί η υποδομή, μιλάμε για χρόνια για να γίνει σωστή υποδομή και η σωστή διαχείριση, ένα σωστό, μια σωστή εγκατάσταση, διαχείριση απορριμμάτων, αποβλήτων. στην αρχή του περσινού έτους τους ρωτήσαμε τι γίνεται, αν έχει προχωρήσει το σχέδιο της εγκατάστασης αυτής και δεν ικανοποιηθήκαμε από την απάντηση των αρμοδίων αρχών, όμως πιστεύω ότι πολλά πράγματα ακόμα πρέπει να γίνουν ε, στην περιφέρεια αυτή. Ε, το βασικό είναι ότι πρέπει να οργανωθεί επιτέλους σωστά ε, η συλλογή των απορριμμάτων αλλά και ο διαχωρισμός των απεριμάτων. Από τη βάση δηλαδή, από τις σκουπιδοντενεκέδες. Ε, αλλιώς δεν θα επιτύχουμε ποτέ μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη λύση. Να αρχίσουμε από, από την αρχή, από το πρώτο βήμα είναι μια περίπτωση παραβίασης των ε, κανόνων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερευνούμε την υπόθεση και ξέρετε ότι το πρόβλημα είναι εξαιρετικά δύσκολο καυτό στην Ιταλία με τα απορρίμματα. Εν συνεχεία, υπάρχουν δύο βασικά λάθη που γίνονται όταν μιλάμε για την αποδοτικότητα των πόρων. Καταρχάς γίνεται μία απλούστευση, ότι προσέχουμε ιδιαίτερα τον τομέα της προμήθειας πρώτων υλών, της εισρωής πρώτων υλών, σαν να είναι αυτό το μόνο πρόβλημα. Και το δεύτερο, όταν μιλάμε για αποδοτικότητα πόρων, αυτομάτως στο μυαλό μας έρχεται ο τομέας της ενέργειας. Αυτό αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ότι χωρίς καμία αμφιβολία Το πολιτικό μήνυμα είναι σαφές στην ανακοίνωση λέμε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα των πόρων ακριβώς όπως το εξηγήσατε εσείς και να μην ασχοληθούμε μονόπλευρα μόνο με το θέμα της προμήθειας των ε, πρώτων υλών. Πιστεύω ότι όλες αυτές οι οικολογικές ε, υπηρεσίες ε, επικρίθηκαν στο παρελθόν ότι δεν χρησιμοποιούνται όσο πρέπει, αλλά αυτό θα διορθωθεί τώρα. Αυτή τη στιγμή η ερώτηση αφορά το Life Plus. Αυτή τη στιγμή δίνουμε μάχη για να το καθιερώσουμε, να το περάσουμε. Εν συνεχεία θα δούμε πώς θα υλοποιηθεί. Είναι μέσα στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών. Εγώ πιστεύω ότι οι δικές μας πολιτικές πρέπει να εφαρμοστούν οριζόντια και στις άλλες βασικές πολιτικές να υπάρχει δηλαδή η διάσταση του Life Plus. 400 Για 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μιλάμε. Αν δείτε το ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το ποσό που δαπανάτε για καθαρά περιβαλλοντικούς στόχους είναι 12,5 δις ευρώ. Είναι μια πολυτέλεια θα έλεγα. Η δυσκολία είναι να πείσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα θέματα περιβάλλοντος. Είμαι βέβαιος ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένους στόχους και ότι το Life Plus θα επιβιώσει και θα υπάρχει, θα, θα, θα, ε, εσωματωθεί στην πολιτική μας. Έχουμε προχωρήσει αρκετά, έχουμε καταφέρει να περάσουν σημαντικές αλλαγές και έχουν αξιολογηθεί αυτές με επιτυχία από περιφέρειες και ε, φορείς σχετικά με τους στόχους τους οποίους πρέπει να θέσουμε. Ποτέ, Ποτέ. δεν θελήσαμε εμείς να ξεκαθαρίσουν ή δεν ήταν μάλλον μια ιδέα αυτή σχετικά με το να είναι συγκεκριμένοι στόχοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς επιθυμούμε πώς να ορίσουμε σωστά τους στόχους. και γι' αυτό η αντίληψη η δική μας νομίζω ότι γίνεται πλέον αποδεκτή. Το ερώτημα που τίθεται είναι θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε προς κάτι το οποίο να είναι απλό με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να χρησιμοποιείται σωστά, να υπάρχουν δεδομένα γύρω από αυτό και σε περιφερειακό επίπεδο και να μπορέσουμε να το εντάξουμε στον κύκλο 2020 να καταστεί θα έλεγα τμήμα των οικονομικών μας πολιτικών σαν στόχος ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες του κοινού. για τις οικονομικές δυσκολίες στην Ευρώπη. και πώς το περιβαλλοντικό θέμα θα λυθεί υπόψη όταν να συζητιούνται τα θέματα τα οικονομικά. Όταν συζητάμε εμείς την έκθεση, την ετήσια για την οικονομική ετήσια ανάπτυξη, η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολύ σοβαρή βέβαια σήμερα πλέον και μετά από την κρίση των χρηματαγορών και με την κρίση του ευρώ. Προσπαθούμε να παραμείνουμε πάντα σημαντικοί εταίροι στα θέματα τα οικονομικά και σε επίπεδο κεφαλαίου αγορών. Κατανοούμε την δυσκολία της κατάστασης αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ότι βρισκόμαστε σήμερα σε μια κατάσταση όπου το περιβάλλον υποβιβάζεται. Έχει μειωθεί η ανάπτυξη του ΑΕΠ και δεν φταίει φυσικά το περιβάλλον για κάτι τέτοιο, για αυτό το οποίο συμβαίνει. το να λέμε ότι το περιβάλλον αυξάνει το κόστος της οικονομικής δραστηριότητας είναι άδικο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει θέμα κόστους, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε το ΑΕΠ να κατεβαίνει και ακριβώς γι' αυτό ε, πρέπει να δούμε τι είδους θέσεις απασχόλησης δημιουργούμε όταν η οικονομική ανάκαμψη υπάρχει και τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε μόνο για το τι θα γίνει με την προστασία του περιβάλλοντος. Το θέμα δεν είναι η ποσοτική ανάπτυξη, αλλά η ποιοτική ανάπτυξη. Όταν λυθεί το πρόβλημα της ποιότητας της ανάπτυξης, τότε θα μπορέσουμε να πετύχουμε πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Δεν πάμε καλά, αλλά δεν πάμε καλά οικονομικά, όχι λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων και πρέπει να λάβουμε υπόψη μα τους παρα, πα, περιβαλλοντικούς παράγοντες για την ανάκαμψη. Marine litter is high on the Commission's agenda. I was myself. Για τα θαλάσσια απορρίμματα είναι ψηλά στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξετίμησα την παρουσία των Ευρωβουλευτών. Um, direction where I intend to follow in the future. So E- είναι ένα θέμα, το θέμα της θαλάσσιας μόλυνσης, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, θα έλεγα, διεθνώς. Αλλά νομίζω ότι υπό το φως των προτάσεων που έχουν γίνει, ήδη από τον Νοέμβριο έχουμε κάποιες κατευθύνσεις. Το σεμινάριο που είχαμε κάνει είναι ότι πλειοψηφία των σκουπιδιών που ε, βρίσκονται στις θάλασσες έρχονται από χερσαίες περιοχές. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει από εκεί το πρόβλημα. Θα πρέπει όλα αυτά τα παραδείγματα να τα λάβουμε υπόψη μας. Σας διαβεβαιώ ότι πρόκειται για μια πολιτική την οποία δεν θα αγνοήσω, δεν θα αναβάλω και είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει άμεσα. Για την Κίνα δεν θα ήθελα να σχολιάσω εδώ, τέθηκε συγκεκριμένη ερώτηση για την πολιτική των Κινέζων. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας δώσω μια γραπτή απάντηση ως προς αυτό. Πάντως οι Κινέζοι θεωρούν ότι έχουν μια ξεκάθαρη πολιτική σχετικά με τη διεθνή τους παρουσία και σκοπεύουν να ακολουθήσουν πολιτικές οι οποίες θα ενισχύσουν τη σημαντική θέση που έχουν στην διεθνή σκηνή. Μέρκες. Πολύ σωστά είπατε για τις πιθανές λύσεις οι οποίες υπάρχουν στα προβλήματα. Σας έθεσα το παράδειγμα της Μισλά όπου δεν πολλούν μόνο τα ελαστικά, αλλά ενοικιάζουν μερικές φορές τα ελαστικά. Στην ουσία πολλούν και τις υπηρεσίες τους μαζί και χρησιμοποιούν τα προϊόντα τους με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Τέθηκαν και άλλες ερωτήσεις για τα πλαστικά απόβλητα και για την Κίνα. Το θέμα είναι όχι τι κάνω, αλλά πώς θα πετύχουμε αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Το δεύτερο γύρος αφορά την βιοπικιλότητα. Ο Γκουσλαφ Σόνικ δεν είναι εδώ. Η Κάρεν ε, Κάντενμπαχ. Biodiversity, βιοπικιλότητα. Σας καλωσορίζω θερμά κύριε Επίτροπε και σας ευχαριστώ που συμμετέχετε και πάλι σε ένα διάλογο με την Επιτροπή μας. Έχουμε τώρα, την, αναφερθήκαμε στην βιοποικιλότητα, την ανάπτυξη και την ποιότητα της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη από μόνη της δεν είναι ο στόχος, μονομερής στόχος, ε, στόχος μας και έχουμε και δύο προγράμματα δράσης το ένα αφορά το, περιβάλλον το έκτο ε, περιβαλλοντικό πρόγραμμα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έληξε το 2010 και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος μα είπε ότι ακόμα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα εκκρεμή και πάρα πολλές ε, δράσεις πρέπει ακόμα να αναλυφθούν. Πολλά πράγματα πρέπει να κάνουμε. Τώρα, σύντομα, θα έρθει η ώρα του 7ου περιβαλλοντικού προγράμματος πότε έχετε πρόθεση να το παρουσιάσετε και με τι τεκμηρίωση, τι άλλα στοιχεία μπορείτε να μας δώσετε. Δεύτερον, έχουμε ανακοινώσει ένα πρόγραμμα ε, δράσεων πρωτοβουλίας. Θα, εσείς ανακοινώσετε μάλλον ένα πρόγραμμα πρωτοβουλίας. Ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτές τις πρωτοβουλίες, ποιοι είναι ενδιαφερόμενοι στη βιομηχανία, στον οικονομικό τομέα, στους πολίτες, ενώσεις κλπ. οργανώσεις. Κύριε Επίτροπε, το 2010 απέτυχε η στρατηγική 2006 της βιοποικιλότητας και είχα χαρεί τότε για τη δουλειά που έκανε η Κομισιόν για την έγκριση του στρατηγικού σχεδίου για το μέλλον του πλανήτου. Ε, έγινε τότε μια σημαντική πρόοδος αλλά ξέρουμε ότι δεν μπορεί να σταματήσουν τα πράγματα εκεί. Η συμφωνία της Ναγκόγιας πρέπει να ακολουθηθεί από άλλα μέτρα. Οι 20 στόχοι που ετέθησαν είναι μεταξύ αυτών και γι' αυτό το Κοινοβούλιο αναμένει με ανυπομονησία τη δημοσίευση της αναπτυξιακής στρατηγικής 2020 που θα μας βοηθήσει και για την αναθεώρηση της ΚΑΠ και της αλληλείας και για τη συνοχή. Με ποιο χρονοδιάγραμμα λοιπόν κύριε Επίτροπε αναμένετε να γίνουν όλα αυτά, τι θα γίνει τους έξι επόμενους μήνες, ποιες νέες μέθοδοι, εργαλεία θα χρησιμοποιήσετε για να εφαρμοστεί πράγματι υπάρχουσα νομοθεσία, ο συντονισμός των προσπαθειών για την προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων θα συμπεριλαμβάνονται στην αυτή στρατηγική. Ευχαριστούμε πολύ. Απαντήσεις του Επιτρόπου. Πέντε λεπτά. Καταρχάς, το 7ο πρόγραμμα περιβάλλοντος. Όπως είπατε σωστά, στο μέσο του έτους θα υπάρξει διαθέσιμη αξιολόγηση του έκτου προγράμματος. Οπότε εκεί θα, τότε θα αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε για να μην, και για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, δεν είμαι αντίθετος με το 7ο πρόγραμμα, ίσα ίσα. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ισχυρά επιχειρήματα και ιδέες. Ε, θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας, βήμα προς βήμα, στα, ζητήματα, στα σημαντικά ζητήματα, να αξιολογήσουμε το έκτο και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Απαντώ ταυτόχρονα και στην ερώτηση της ε, Σαντρίν γιατί μας ρώτησε, με ρώτησε τι θα κάνουμε, τι σχεδιάζουμε για το επόμενο έτος. Πολλά εξαρτώνται από τις αποφάσεις που θα πάρουμε το 2011. Ε, γεωργική πολιτική, αλλιευτική, πολιτική συνοχής κλπ. Έχουμε τις δικές μας προτάσεις στη στρατηγική βιοπικιλότητας, άλλες προτάσεις για την αποδοτικότητα των πόρων και η έκθεση αξιολόγησης ε, της έκτης ε, ε, έκθεσης περιβάλλοντος. Πρέπει να δούμε όλες αυτές τις αξιολογίες και τις εκθέσεις γιατί ο κόσμος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα και πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα νέα στοιχεία όταν πριν από 10 χρόνια μιλούσαμε για το έκτο περιβαλλοντικό πρόγραμμα, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Ε, απαντώ λοιπόν ότι μάλλον στις αρχές του επόμενου έτους, ε, του 2012, θα παρουσιαστεί η συνέχιση του έκτου περιβαλλοντικού προγράμματος, ίσως με τον τίτλο «Έβδομο περιβαλλοντικό πρόγραμμα». Έχουμε δηλαδή, ε, πρέπει να έχουμε καιρό, χρόνο μπροστά μας να αξιολογήσουμε αυτά τα οποία έχουν συμβεί εντωμεταξύ μεταξύ και τις αλλαγές. Χωρίς ε, βεβαίως να χάσουμε και πολύτιμο χρόνο φέτος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε όλοι και να μην χάσουμε καμία ευκαιρία δημοσιονομικές προτάσεις θα υπάρχουν στο τραπέζι και θα ε, καλύπτουν τα επόμενα 5-10 χρόνια. όταν θα έχουν ληφθεί οι αποφάσεις οι δημοσιονομικές θα είναι πια πολύ αργά να παρουσιαστεί το 7ο περιβαλλοντικό πρόγραμμα πρώτα. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν οι οικονομικές αποφάσεις ε, και μετά να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα. Αλλά παρακαλώ μην, παρανοείστε ότι εγώ θέλω να κολυσιεργήσω ή να καθυστερήσω γιατί πολλές φορές με κατηγορούν γι' αυτό καθόλου. Ε, ε, για τη μελέτη επιπτώσεων ε, ασχολούνται εσωτερικές υπηρεσίες της Κομισιόν ε, και σε μερικές εβδομάδες θα ολοκληρωθεί η μελέτη επιπτώσεων. Είμαστε στην τελευταία φάση. Ε, έχουμε επίσης και έναν κατάλογο υποστόχων παράπλευρων στόχων, όπως παραδείγματος χάρη την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και άλλα συναφή θέματα. Βασικά δηλαδή πιστεύω ότι απάντησα και στην ερώτηση της Αντρίν και κάτι ακόμα τελευταίο. Η υπάρχουσα νομοθεσία Natura, γιατί το Natura 2000 είναι στη φάση της υλοποίησης. Έχουμε τώρα, το έχουμε αυξήσει, διευρύνει από 70 σε 80%. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα σωστά προγράμματα διαχείρισης ε, υπάρχουν και είναι ε, έτοιμα να εφαρμοστούν και πρέπει να παρακολουθούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή του Natura. Ευχαριστώ. Το τρίτος γύρος αφορά την υλοποίηση, την εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας. Και αρχούμε με τον κύριο Φλόρενς που μόλις έφυγε, ξαφανίστηκε και προχωρούμε, προχωρούμε τον Ντάν Γιούργενσον. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Εξαιρετικές οι απαντήσεις σας ως συνήθως. Να θέσω κάποιες ερωτήσεις για τα εντομοκτώνα, για τον κανονισμό για τα εντομοκτώνα. Εδώ και λίγα χρόνια υιοθετήσαμε ένα νέο κανονισμό σχετικά με την εμπορία των προϊόντων αυτών και κανονικά θα πρέπει τον μήνα Ιούνιο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και πρέπει να έχει επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα κατάλογο για τα απαραίτητα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται στα προϊόντα αυτά. Οι υπάρχουσες απαιτήσει καθορίστηκαν το 1991 για τα και από τότε έχει αλλάξει η νομοθεσία και απαιτούνται να υπάρξουν νέες απαιτήσεις. Έχετε εσείς πληροφορίες για το αν θα μπορέσετε να ξεκαθαρίσετε τις απαιτήσεις σας τον Ιούνιο. Και αν όχι, τι κάνετε για να επιταχύνετε τη διαδικασία. Και μια συμπληρωματική ερώτηση. Δεν έχει καμία σχέση με τα ζυζανιοκτώνα, αλλά για τα υπόλοιπα των χημικών ουσιών στα τρόφιμα. Πολλές φορές όταν ελέγχουμε λαχανικά και οπόρες στα ε, καταστήματα βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζονται σωστά οι κανόνες και υπάρχουν ίχνοι στοιχείων. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ λέει ο κύριος Φλόρενς. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, θα πρέπει επιτέλους να ε, κοιτάξουμε την εφαρμογή ε, των αποφάσεων και των ε, νομοθετικών κανόνων. Είναι πολύ λυπηρό αυτό το φαινόμενο ότι λαμβάνουμε και εγκρίνουμε αποφάσεις και συνεχεία δεν εφαρμόζονται. Θα ήθελα σας παρακαλέσω κύριε Επίτροπε, να υψώσετε τη φωνή σας και να, ε, ώστε να, και να φέρετε τους ε, παραβάτες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τώρα τα ε, παρασιτοκτόνα, δεν καταλαβαίνω γιατί η Κομισιόν δεν χρησιμοποιεί την αρχή της πρόληψης όσον, όσον αφορά τα ζυζανιοκτώνα και τις μέλισσες, τη μελισσοκομεία. Έχουμε περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά σε ορισμένα κράτη-μέλη λείπει τελείω το πλαίσιο ελέγχου και επιθεώρησης. Τώρα, ε, πριν από μερικά χρόνια είχε συσταθεί μία επιτροπή για να δημιουργηθεί ένα σώμα επιθεωρητών ελεγκτών και είχαμε προτείνει τότε όλα αυτά να περάσουν στην κοινοτική νομοθεσία. Ε, υπάρχουν τεράστιες διαφορές, διότι σε πολλές χώρες δεν υπάρχει καμία συστηματική, συστηματικός έλεγχος όλων, της εφαρμογής όλων αυτών των περιβαλλοντικών ε, κανόνων, ενώ σε άλλες χώρες υπάρχουν τακτικές ε, τακτική έλεγχη. Θα κάνετε τίποτα έτσι να εφαρμοστεί ένα συντονισμένο πλαίσιο ελέγχων. Ευχαριστώ η, κυρία Χάσλ, Ένα από τα θέματα της νομοθεσίας που μας ε, αφορά είναι τα ε, καύσιμα τα που χρησιμοποιούνται για την αυσιπλοεία. Είχα, μας είχατε υποσχεθεί ε, την, το την εφαρμοστική νομοθεσία πέρσι αλλά μέχρι φέτος δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό το θέμα ε, αφορά την υγεία των πολιτών μας και επίσης περιμένουμε την οδηγία των εθνικών ορίων εκπομπών, τα εθνικά όρια εκπομπών. Ε, και πάλι εδώ δεν έχουμε τίποτα. Είχαμε συζητήσει πέρσι έντονα την ε, ατμοσφαιρική πολιτική και όλα τα συναφή θέματα Πού βρισκόμαστε τώρα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Οι ιδιοκτήτες ε, των ε, ferry boats της Βαλτικής βρίσκονται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε πιστεύω θα ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα καύσιμα που χρησιμοποιούν και τη συναφή νομοθεσία. Τα ερωτήματα που αφορούν τα ζυζανιοκτώνα ή παρασιτοκτώνα δεν έχω απάντηση αλλά θα φροντίσω να σας δοθούν γραπτές απαντήσεις όσο το δυνατόν συντομότερο. Δεν νομίζω, δεν έχω μάθει ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις. Ελπίζω, φαντάζομαι ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά δεν γνωρίζω συγκεκριμένα τι ισχύει για αυτές τις απαιτήσει του κανονισμού. Δεν αναμένουμε πάντως κανένα πρόβλημα στην εφαρμογή του. Αλλά σας είπα και το ξαναλέω θα λάβετε γραπτή απάντηση. Γενικά το θέμα της εφαρμογής είναι πολύ σοβαρό. Και δεν υπάρχει καμία πανάκια έτοιμη πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Γιατί υπάρχουν νομοθετήματα που δεν μπορούν να συνδυαστούν εύκολα σε όλη την Ένωση. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή πολιτική συζήτηση για αυτό το πρόβλημα και σχεδιάζω να κάνω μια πολιτική ανακοίνωση κατά τα μέσα του έτους όπου όλα αυτά τα θέματα που θίξατε όπως σωστά κριτήρια επιτήρησης ή ελέγχου ή καμιά ειδική οδηγία ή μία υπηρεσία εφαρμογής της οδηγίας για τα απόβλητα σε πανενωσιακό επίπεδο και τέτοια. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε με τρόπο πιο συστηματικό σε επίπεδο συστήματος. Και Αυτό θα το φροντίσουμε στο δεύτερο ήμιση του έτους. Θα σας δώσω ένα πολιτικό έγγραφο όπου πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα για να μην μείνει τίποτα που να μην έχει εξεταστεί. Κάτι άλλο που βλέπω να έρχεται είναι ότι θα ξέρετε ότι ήμουν επικεφαλής της ε, ομάδας διαπραγμάτευσης, ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Σλοβενία, για τη Σλοβενία. Και Είχαμε δει τότε ότι στα απόβλητα και στη διαχείριση των αποβλήτων υδάτων χρειάζονται, χρειάζεται πολύ σημαντική επένδυση. Επένδυση λέγω. Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε την ενωσιακή νομοθεσία. Και ακριβώς κατά τη διάρκεια της θητείας μου θα εκπνεύσει η μεταβατική περίοδος είναι λοιπόν πολύ σημαντικό όταν και εμείς και εσείς θα μιλήσουμε για το μέλλον της πολιτικής συνοχής να το λάβετε υπόψη σας ε, διότι δεν υπάρχει τρόπος οι νέες αυτές χώρες μέλη να μπορέσουν μόνες τους να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Θα είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό να μην το ξεχάσουμε. Είναι εξάλλου και πολύ λογικό να συγχρηματοδοτηθεί σε ενωσιακό επίπεδο η προσπάθεια αυτή γιατί δεν βοηθάει μόνο τις συγκεκριμένες χώρες μέλη αλλά όλους και όλες. Παραδείγματο χάρη η μόλυνση του Δούναβη δεν είχε προβλεφθεί, δεν σε τέτοιο επίπεδο τουλάχιστον. Όσο για το θείο και το διοξίδιο ή οξίδιο του, δεν ήξερα πριν, αλλά τώρα ξέρω ότι πρόκειται να, σε ένα-δυο μήνες να έρθει πρόταση γι' αυτό. Το συζητήσαμε και όταν λέγαμε για την ποιότητα του αέρος, διότι ακριβώς σε αυτό βασιστήκαμε, να γνωρίζουν όλοι οι επίτροποι το πρόβλημα. Δύο βασικά θέματα βλέπουμε εμείς. Σε συγκεκριμένους τομείς όπως ορισμένα μόρια ή αιωρούμενα στοιχεία το όζων βλέπουμε να υπάρχουν προβλήματα. Και αυτό είναι πρόβλημα της πηγής που τα εκπέμπει, που είναι κυρίως οι μεταφορές το πρόβλημα λοιπόν δεν θα λυθεί αν απλώς βάλουμε όρια στην οδηγία. Πρέπει να δούμε και ποιος δημιουργεί αυτά τα σωματίδια. Πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι οι πραγματικές προτάσεις στους τομείς των συναδέλφων μου θα έχουν αποτέλεσμα και τα κράτη-μέλη θα δουν διαφορά. Αυτό συζητήσαμε για την ποιότητα του αέρα. Πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι ανάλογο με αυτό που είχαμε κάνει για τις κλιματολογικές αλλαγές και την ενέργεια. Δηλαδή πολιτική μεταφορών συν περιβάλλον για να λυθεί το πρόβλημα του αέρα. Το αργότερο μέχρι το, δεκα... το τέλος του 2013 αυτό να μην το θεωρήσετε καθυστέρηση ή αναβολή. Αντίθετα, η οδηγία ΝΕΚ θα έρθει σύντομα σε συζήτηση και το βασικό πρόβλημα είναι τι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα, θα υποστηριχθεί όπως πρέπει από τα προγράμματα που, για τα οποία είναι υπεύθυνοι οι συνάδελφοί μου, ώστε όμως να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίος γύρος διάφορα εννέα βουλευτές ζήτησαν το λόγο. Ένα λεπτό όμως ο καθής. κάνουν πρώτον. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Καταρχήν, σας συγχαίρω για όσα έχετε κάνει για το θέμα της αυταρκίας. Αναφέρατε σαφείς στόχους. Μέχρι το 2050 θα μπορούσαμε να έχουμε λύσει το πρόβλημα των μη ανανεώσιμων πηγών και της προστασίας της βιοπικιλότητας. Έχω λοιπόν τρία ερωτήματα. Πρώτον, τι σκοπεύετε να κάνετε για το GPI και τις εταιρικές αίσεις καινοτομίας για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δεύτερον, τι σχέση έχει αυτό με τις πρωτοβουλίες για τις πρώτες ύλες και τρίτον, για τις νομικές διευθετήσεις, τι στόχους έχετε θέσει για τις εκπομπές. Ευχαριστώ, τελειώσατε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, είπα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Επίτροπο, τον συγχαίρω για την καλή δουλειά που έκανε μέχρι τώρα. Η ερώτησή μου αφορά τη συμφωνία. We and based on the assessment that uh, has been uh, done for the Commission, it was... Έχουν γίνει ορισμένες εκτιμήσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φαίνεται ότι 480 εκατομμύρια εκτάρια δάσους θα καταστραφούν μέσα από τη συμφωνία αυτή. Το 11% δηλαδή των ε, τροπικών δασών της Βραζιλίας. Και δεν μιλάω εδώ για τη μετακίνηση ε, των ε, πληθυσμών που θα αναγκαστούν να φύγουν για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Συνειδητοποιείτε το μέγεθος του προβλήματος και παίρνετε μέρος στις συζητήσεις αυτές ε, για τα δάση. Τι ε, επιπτώσεις έχουν οι αποφάσεις της Ναγκόγια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο ερωτήματα λέει ο κύριος Κράμερ. Το πρώτο αφορά τις ε, εκπομπές βιομηχανικών μονάδων. Είχαμε εγκρίνει έναν κανονισμό πέρσι αλλά ήδη υπήρχαν νέες ομάδες εργασίας για, μια, για ένα νέο κανονισμό των ε, βιομηχανικών εκπομπών, βλαβερών εκπομπών. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι η Κομισιόν έχει αναστείλει τις ε, εργασίες αυτού του θέματος. Ήθελα να, να σας ρωτήσω αν ξέρετε τους λόγους και αν αυτό ισχύει ή αν κάνω λάθος. Δεύτερον, στο πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν ε, μακροπρόθεσμα λέει ότι Α, ότι στα βαρέα φορτηγά θα ασχοληθεί η Κομισιόν με τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και θέλω να ρωτήσω, ε, προβλέπεται η Κομισιόν να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση στα ε, αυτοκίνητα. Ο Νοέμβριο η ΕΦΣΑ Κύριος Έγγραφο κατευθύνσεων σχετικά με την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών μαζί με μια γνωμοδότηση σχετικά με τις επιπτώσεις τους σε μη στοχευόμενους οργανισμούς. Το 2011 η Επιτροπή θα προσιάσει μια πρόταση για αυτές τις περιβαλλοντικές κατευθυντήριες γραμμές που θα λάβουν κανονιστική ισχύ μέσω Comitology και θα αποτελέσουν τη βάση για τις αιτήσει αδειοδότησης γενετρικά τροποποιημένων καλλιεργιών. Δεδομένου ότι η πρόταση είναι σαφώς σχετική με περιβαλλοντικά θέματα. Μπορείτε να μας ενημερώσετε με ποιον τρόπο έχετε εσείς και ε, η Γενική Διεύθυνση ΕΜΒΗ, πώς έχετε εμπλακεί στη διαδικασία μέχρι σήμερα. Θα βεβαιώσετε με τις πράξεις σας ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες λαμβάνονται επαρκώς υπόψη. Τι γνώμη έχετε τέλος για τις τέσσερις ποικιλίε γενικά τροποποιημένων οργανισμών που ετοιμάζει να εισάγει στην αγορά ο συνάδελφός σας επίτροπος κ. Ντάλι, ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαβουλεύσεις για την ανάλυση ρίσκου. Ο uh, Oreste Rossi. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, γνωρίζετε ότι για το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για το 2011 αναφέρεται και το θέμα της πολιτικής προστασίας. Τι θέλετε να πετύχετε στον τομέα αυτό, θέλετε να υπάρξει ένα συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις κατεπίγουσες παρεμβάσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν καταστροφές σε πολλές χώρες, πλημμύρες ας πούμε ποταμών που διασχίζουν περισσότερες χώρες ή σεισμοί κτλ. Αυτό θα μπορούσε να είναι πιθανό μετά από τις συνέπειες που έχει στην, στο κλίμα ε, ή μάλλον τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω των κλιματολογικών αλλαγών ή θέλετε να δημιουργήσετε ένα ταμείο για άμεσες παρεμβάσεις το οποίο να είναι άμεσα διαθέσιμο. Ε, υπάρχει ένα τέτοιο ταμείο σήμερα το οποίο ενεργοποιείται όμως μόνο αν οι ζημίες είναι ιδιαίτερα υψηλές, σχεδόν ποτέ δηλαδή. Αν όμως υπάρχει ένα ταμείο το οποίο είναι εύκολα διαχειρίσιμο σε έφθετο χρόνο, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο και για το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Η κυρία Γεώργεβα είναι υπεύθυνη για τα θέματα της αστικής προστασίας. Γιάννος Άντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από εννέα μήνες περίπου το Κοινοβούλιο υιοθέτησε το ψήφισμα για την απαγόρευση ορισμένων τεχνολογιών εξόριξης άνθρακα. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή πώς έχει προχωρήσει ε, αυτό το θέμα. Δεύτερον, σας στείλαμε μία πρόταση σχετική με την εισαγωγή ενός ε, περιβαλλοντικού τέλους εισφοράς στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε λάβει υπόψη αυτή την πρόταση, αν την υποστηρίζετε, έτσι ώστε οι συνάδελφοί μου μπορούν να αρχίσουν τις τεχνικές διαβουλεύσεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι ο Επίτροπος είναι αρμόδιος για τη μείωση των επιδοτήσεων διοξιδίου του άνθρακα. Δίνω το λόγο στην επόμενη ομιλήτρια, κυρία Κλάς. Ευχαριστώ ε, κύριε Επίτροπε. Θέλουμε όλα να τα συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται. Τέθηκε το ερώτημα του πώς μπορούμε να μετρήσουμε την ποιότητα της ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία πρόταση για, την, ε, για έναν κανονισμό που θα καλύπτει όλα τα θέματα περιβάλλοντος, ισολογισμός δηλαδή. Και αναρωτιέμαι αν μια τέτοια γραφειοκρατία, ένα τέτοιο γραφειοκρατικό άχθος είναι βιώσιμο. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια. Αφού δεν έχουμε τις ε, παραμέτρους μέτρησης ε, δημιουργούμε μία ε, τεράστια γραφειοκρατία υποτίθεται για να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα αλλά δεν νομίζω να επιτύχουμε. Εγώ λέει ο πρόεδρος, είμαι εισηγητής αυτού του ντοσιέ και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ αποδοτική αυτή η εργασία, διότι η UNEP θα, είχε, θα ήθελε πάρα πολύ να έχει αυτά τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία εγώ θα επεξεργαστώ πολλά ερωτήματα λοιπόν κύριε Επίτροπε και ό,τι δεν μπορείτε να απαντήσετε θα το λάβουμε γραπτός. Έχετε το λόγο. Ναι, ναι, δυστυχώς λέει ο κύριος Επίτροπος. Joint, uh, the question which uh, Sir asked, uh, joint technology initiatives and... Οι πρωτοβουλίες, οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες και οι εταιρικέ συνεργασίες ε, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Εγώ πιστεύω ότι και οι δύο αυτές ιδέες έχουν συζητηθεί στο παρελθόν και πιστεύω σε αυτές. Τα είχαμε πει και στο σεμινάριο για τους καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης. Έχουμε περιορισμένους πλέον πόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τη μία και από την άλλη έχουμε αυξανόμενες ανάγκες οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καλύτερος τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα που έχουμε τα χρήματα αυτά είναι η μόχλευση είτε μέσω συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή ευρωπαϊκά χρήματα ναι. συν-ιδιωτικά, συν-εθνικά, να υπάρξει δηλαδή μια εταιρική σχέση και με τον ιδιωτικό τομέα και ακριβώς ε, τέτοιες ιδέες εφαρμόζονται στα πλαίσια των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλειών. Θεωρούμε ότι τα μέσα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για το περιβάλλον γενικότερα. Φυσικά. Καινοτόμα μέσα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, κατά προτίμηση στο περιβάλλον. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ε, σκεφτόμαστε επίσης να προχωρήσουμε σε εταιρικέ συνεργασίες και στον τομέα της έρευνας και της αναζήτησης της καινοτομίας. Τώρα η πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλε. Έχει υπάρξει μια αναβολή. Κανονικά έπρεπε να ψηφιστεί αύριο, αλλά θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Ένα από τους, ένας από τους τρεις πυλώνες αφορά την αποτελεσματικότητα των πόρων και τη σχέση του θέματος με το περιβάλλον. Νομίζω ότι καλύπτεται γενικά στην περίπτωση αυτή ε, το θέμα του περιβάλλοντος. Τώρα για τη συμφωνία Μερκοσούρ, στην οποία αν κατάλαβα καλά αναφερθήκατε. Δεν έχω ακούσει τα, τους αριθμούς τους οποίους αναφερθήκατε. Θα τα εξετάσω και προφανώς αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συζητιούνται έτσι κι αλλιώς τα θέματα πριν καταλήξουμε σε λήψεις αποφάσεων. Αυτό το οποίο μπορώ να κάνω είναι να εξετάσω το θέμα πιο συγκεκριμένα, να ενημερωθώ καλύτερα και να δω ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της ε, προσπάθειας η οποία γίνεται στη Βραζιλία και στα πλαίσια των κανονισμών που έχουν υιοθετηθεί πρόσφατα για την εκμετάλλευση των εισαγόμενων μάλλον προϊόντων ξυλίας. Προχωράμε επίσης στην σύναψη συμφωνιών σε εθελοντική βάση για τα προϊόντα αυτά, την παραγωγή και την εμπορία τους με συγκεκριμένες χώρες. για τα ETS. Δεν ξέρω να σας δώσω στοιχεία, αλλά το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω ήταν ε, η πρώτη αφορούσε τα ETS, η δεύτερη τα γενετικά τροποποιημένα και η τρίτη την πολιτική προστασία. Και τα τρία είναι εκτός χαρτοφυλακίου μου, αλλά θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση. Λοιπόν, τα ETS, δεν ξέρω ακριβώ που είμαστε τώρα. Εμείς ενεπλάκημεν στη συζήτηση αυτή μόνο όταν φτάσει αυτό το θέμα σε γραφείο επιτρόπου. Πριν από αυτό η εμπλοκή μου σε τέτοιου είδους δραστηριότητες δυστυχώς ε, δεν είναι η συμμετοχή μου καθοριστική για τα γενετικά τροποποιημένα. Η διαδικασία την οποία ακολουθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προβλέπει την στενή συνεργασία πριν από την αδειοδότηση τέτοιων ουσιών και σε επίπεδο περιβάλλοντος κοιτάμε τις πιθανές συνέπειες και ταυτόχρονα ο Επίτροπος Ντάλη στην ουσία έχει κληρονομήσει μια πλήρη ομάδα από την προηγούμενη μου σε εισαγωγικά δουλειά που εξετάζουμε τις πιθανές επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων. Βρισκόμαστε λοιπόν σε φάση εργασίας από πλευρά του αρμόδιου επιτρόπου. Για την πολιτική προστασία. Ξέρω αρκετά γύρω από το θέμα αυτό. Είχα εμπλακεί κι εγώ παλιότερα. Η Κρυσταλίνα, η συνάδελφος, θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστούν κάποιες νέες ιδέες και να ενθαρρυνθεί μια κάποια συζήτηση. Το Ταμείο Αλληλεγγύης δεν έχει την χρησιμότητα, δεν προβλέπεται να έχει τη χρησιμότητα της άμεσης διαθεσιμότητας και αντίδρασης προς τα κράτη-μέλη. Μεσολαβεί μια ολόκληρη διαδικασία σχετικά με όρια, κριτήρια κτλ. Και θα πρέπει να υπάρξει έγκριση των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η οικονομική βοήθεια περίπου κάνει ένα χρόνο να φτάσει. Η πολιτική προστασία είναι άμεση βέβαια και παρέχεται άμεσα, αλλά αυτό είναι διαφορετικό θέμα. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς και οικονομικά, όχι μόνο πρακτικά, να αντιδράσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο ελείπει και αυτό είναι κάτι το οποίο η συνάδελφός μου θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει. Κύριε Ρέντερ, θα σας δώσω γραπτά Τις τελευταίες εξελίξεις και τέλος το ερώτημα του πέραν του ΑΕΠ αν πιστεύει κανείς ότι τα δεδομένα για το ΑΕΠ ε, συλλέγονται εύκολα, κάνει λάθος. Το ΑΕΠ σήμερα είναι θα έλεγα μια πηξίδα μέσω της οποίας μπορούμε να γνωρίζουμε την ταχύτητα της λειτουργίας της μηχανής χωρίς όμως να γνωρίζουμε σε ποια κατεύθυνση πηγαίνουμε και πόσα κάψιμα έχουμε. Αυτό είναι το θέμα λοιπόν και γι' αυτό θα πρέπει όλοι να λάβουμε υπόψη μας το πώς εξελίσσονται τα πράγματα εξεπλάγην ακούγοντας ότι η Επιτροπή σας σήμερα το πρωί δεν έκρινε θετικά την έκθεση για τα πέραν το ΑΕΠ, των πέραν του ΑΕΠ παραγόντων. Νομίζω ότι σήμερα έχουμε περισσότερες ερωτήσεις από ότι απαντήσεις, αλλά παρακαλώ με την πηξίδα και τις κατευθύνσεις που ακολουθούμε σήμερα κάνουμε λάθος δεν πηγαίνουμε σε σωστές κατευθύνσεις και αν συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια λάθη τότε το πρόβλημα θα είναι μεγάλο. Ευχαριστώ Γιάννη Σποτότσκι, όπως πάντα ήσασταν ιδιαίτερα επεξηγηματικός, πρόθυμος. Ξέρουμε ότι δίνετε μάχες σε πάρα πολλά θέματα. Είδα σημειωμένα 73 θέματα να έχετε σημειώσει στα έγγραφά σας. θα ήθελα να πω λέγοντας ότι το 2011 είναι μια πολύ αποφασιστική χρονιά στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Θα αποφασίσουμε για πολλά θέματα φέτος όπως η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, της αλλιευτικής πολιτικής των διαφορετικών ταμείων και όλα τα άλλα πολλά σημαντικά θέματα τα οποία έχετε αναλάβει. Νομίζω ότι θα συνεργαστούμε και να ορίσουμε σωστότερα την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Cross portfolio uh, deliberations. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα στην επόμενη ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ελπίζω μια συζήτηση σαν τη να μην καθυστερήσει.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 So, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε τώρα. Τρει ψηφοφορίε έχουμε. 22. Äh, Είμαστε στο, στο σημείο 22 της ημερήσιας διάταξης, έκθεση 2010 για ναι. την εφαρμογή της ε, πολιτικής ε, συνοχής των προγραμμάτων πολιτικής ε, συνοχής 2007-2013, ε, εισηγητής Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες και αρχίζουμε με την ψηφοφορία τροπολογία 2 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Κατά, άποχες, δεκτή. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η, τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 4, υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Επτά, Τοπολογία επτά υπέρ. Κατά, Άποχες. Απορρίπτεται. 8. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. 9. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. 10. Υπέρ. Κατά. Δεν ψήφισε το ΕΛΚ. Αποχές. Ξανά, ξανά. Τη 10, τροπολογία 10, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 11, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 13, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 και 21 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή, δεκτές. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Άποχες Α, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Αμέσως. ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία Λίγο. Ε, ε, πέρας της ψηφοφορίας 51 ψήφι υπέρ μία αποχή, μία ψήφος κατά. Συγχαίρω λοιπόν τον εισηγητή Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες. Επόμενο θέμα, σημείο 23 Also 23. Πολιτικές προκλήσεις και δημοσιονομική πόρη για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013. Συντάκτη γνωμοδότησης Γκέρμπεν Γιάν Γκερμπράντι. Είχαμε μια πρώτη πρόταση που δεν είχε καλύψει όλους εάν μπορούμε να την ψηφίσουμε ε, έτσι ή αν δεν γίνεται να ψηφιστεί η κοινή τροπολογία 1. Α, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Λοιπόν, να ψηφιστεί ως έχει το joint, το, τροπολογία, κοινή τροπολογία 1. 1. Υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ την πρώτη τροπολογία, τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε, πέρασε τη ψηφοφορια Ε, ίσα ίσα, εγκρίνεται, εγκρίνεται 28 υπέρ 26 κατά. Προχωρούμε. Στην παράγραφο 1 είναι το αρχικό κείμενο. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ για τροπολογία 2. Έληξε ψηφοφορία. Δεκτή. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 12. Καταπίπτει. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 8. Υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή εννέα υπέρ κατά αποχές δεκτή δέκα σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 14. Υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. Προχωρούμε τροπολογία 20. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 19. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 32 Α, καταπίπτει. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 34 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 34 παρακαλώ. Έληξε η ψηφοφορία. Δεκτή. 35 υπέρ. Ναι κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 37 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 38 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 39 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 43 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ωραία. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. 55 υπέρ, 2 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Θερμά συγχαρητήρια κύριε ερμπράντι για αυτή την ε, γνωμοδότηση. Και η τελευταία ψηφοφορία σήμερα. Αδιαδικαστικό, Πρόεδρε. Ζητώ να αφαιρεθεί το θέμα από την ημερήσια διάταξη και να αποφασίσουν να το συζητήσουν οι συντονιστές αύριο διότι η Επιτροπή Δημοσίας Υγείας έχει ως καθήκον να θέσει κριτήρια για να διασφαλίσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας και αντί για αυτό εδώ ο συγκητής μας ζητάει να επιλέξουμε τεχνολογίες ανταγωνιστικές μεταξύ τους οι δε έρευνες της Κομισιόν δείχνουν ότι οι εκπομπές και από τις δύο αυτές τεχνολογίες μπορούν να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία ότι το πέρασμα των ακτίνων αυτών από το σώμα μπορεί να βλάψει το σώμα σοβαρά. Δηλαδή στην ουσία απλώς προωθούμε έναν κατασκευαστή έναντι άλλου και του δίνουμε ένα εμπορικό προνόμιο ενώ μπορεί και μπορεί αυτό το προνόμιο να είναι πολύ σημαντικό γιατί χιλιάδες τέτοιων μηχανών θα εγκατασταθούν. Δεν έχουμε πραγματικά εγγεγραμμένα τα συμφέροντα που εκτίθενται εδώ ή που κρύβονται εδώ και μπορεί κάλλιστα να πρόκειται για κρυμμένα εμπορικά συμφέροντα. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε την αρχή της ψηφοφορίας αυτής. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Είμαστε στο παραπέντε της ψηφοφορίας και η Επιτροπή είναι ελεύθερη να αποφασίσει και να κάνει αυτό που θέλει εάν δεν ψηφίσουμε δεν θα εξαφανιστεί το θέμα αυτό στην Ευρώπη. Ε, βλέπω ότι στην αγορά παρουσιάζονται συνεχώς καινούργια προϊόντα, καινούργιες καινοτομίες. Ελπίζω αυτά να έχουν καλυφθεί από τις τροπολογίες έτσι όπως πρέπει να το κάνει η Επιτροπή μας. Εμείς δεν είμαστε η Διευθύνουσα Επιτροπή, απλώς γνωμοδοτούμε. Η αρμόδια επιτροπή δεν είμαστε εμείς. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο να το αναβάλουμε. Έχουμε τροπολογίες, έχουμε τον συντάκτης γνωμοδότησης, έχουμε ολοκληρώσει όλη τη διαδικασία. Εγώ είμαι υπέρ της ψηφοφορίας. Θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε ίσως το διαδικαστικό του κυρίου Ντέιβις. Θα ρωτώ λοιπόν, ο Ρίχαρτ Ζέμπερ έχει κάτι να μας πει, πρόεδρε. Θα ήθελα να ξέρω εάν αναβάλουμε προλάβει την ολοκλήρωση της διαδικασίας η, η αρμόδια επιτροπή. Θα πρέπει και η επικεφαλής, η αρμόδια επιτροπή επί του θέματος να λάβει γνώση της αναβολής μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι στην Επιτροπή Μεταφορών που είναι η αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή και παρακολουθώ τα θέματα αυτά στο σκιώδη συγγήτρια. Νομίζω ότι δεν υπάρξουν συνθήκες οι οποίες ε, ε, θα οδηγήσουν στην αναβολή ή πρέπει να οδηγήσουν στην αναβολή. Έχετε δίκιο κύριε Πρόεδρε λέγεται, λέγοντας ότι υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες και θα αποφασίσουμε πάνω σε αυτές αυτά τα οποία είπε ο πολύ καλός συνάδελφος Chris Davis για τα εμπορικά συμφέροντα κτλ. Εμείς δεν ε, ε, υποδεικνύουμε ή δεν επιβάλλουμε ποιος θα επιλεγεί και ποια τεχνολογία θα επιλεγεί. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δουν τι συμβαίνει στα αεροδρόμια, στις αεροπορικές εταιρείες και στις εθνικές υπηρεσίες, να δουν τι υλικό είναι διαθέσιμο και ανάλογα να πάρουν τις αποφάσεις τους. Δεν υπάρχει λόγος να μην προχωρήσουμε λοιπόν. Αγιάλα Σέντερ και μετά θα κάνουμε την πρόταση. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ συμφωνώ με την κυρία Φώστερ. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε αυτήν την γνωμοδότηση η οποία είναι γνωμοδότηση προς την αρμόδια επιτροπή, την Επιτροπή Μεταφορών. Ζητάμε εμείς ε, να προωθηθεί ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί αρκετά στην ομάδα, στις ομάδες. Η πρόταση είναι αρκετά ανοιχτή και δεκτική δεν υπάρχει κάτι το διφορούμενο, απλά λέγει ότι ε, πρέπει να δούμε ε, ποιες είναι οι διαθέσιμες τεχνολογίες σήμερα. Να επιλεγεί ζητάει το Κοινοβούλιο η τεχνολογία η οποία παρουσιάζει τους μικρότερους κινδύνους ε, για την ανθρώπινη υγεία, για το σεβασμό της, του απορρίτου, της εμπιστευτικότητας η Ευρώπη θα πρέπει να επιλέξει για το μέλλον την τεχνολογία η οποία να επηρεάζει το λιγότερο δυνατόν την υγεία των φυσικών προσώπων. Νομίζω ότι η πρόταση αυτή είναι ιδιαίτερα ρεαλιστική και θα πρέπει παρακαλώ να ψηφίσουμε τώρα. Ο Chris Davis έκανε πρόταση αναβολής της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε ποιος είναι υπέρ της αναβολής. Κατά. Αποχές. Είναι σαφής η πλειοψηφία υπέρ της διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Και προχωρούμε. Ε, τροπολογία 1. Κρίς Ντέιβις. Ποιος είναι υπέρ. Κα, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Επίσης του Κρίς Ντέιβις. Υπέρ. Κατά. Ένα λεπτό. Βιάστηκα, λέει ο πρόεδρο. Πρώτο τμήμα της τροπολογίας 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Α, το δεύτερο τμήμα παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά. Της τροπολογίας 8. Έληξε ψηφοφορία. Ναι, δεκτό το δεύτερο, το δεύτερο μέρος. Δεν δούλεψε το μηχάνημα της κυρίας Αγιάλα, αλλά δεν νομίζω να είχε και επίπτωση στο αποτέλεσμα. Τροπολογία 7, πρώτο τμήμα, υπέρ κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, εποχές, δεκτό. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι. Τροπολογία 10. Υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. Τροπολογία 11. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές check. Ηλεκτρονικά παρακαλώ την 5. Έληξε η ψηφοφορία. Απερίφθη, απερίφθη. Τροπολογία 6, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά παρακαλώ τη 15 έληξε έγινε δεκτή 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τα υπόλοιπα καταπίπτουν. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Το 21, ναι. 21. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παρα, ε, τροπολογία 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ Α, καταπίπτει 25. 29, 29, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 καταπίπτει. 31 Chris Davis υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 35 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 36 καταπίπτει, 37 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή 44 υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. 45 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 46 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 47 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 48 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 49. Ε, ηλεκτρονι... Α, τη 48 παρακαλώ, ηλεκτρονικά. 48. Έληξε τη ψηφοφορία. Δεκτή. Ε, Έχουμε 62 στην αίθουσα και 58 ψήφισαν. Τέσσερις δεν έλαβαν μέρος. Δεκτή λοιπόν. Δεκτή λέει ο πρόεδρος. 49. Υπέρ. Ε, ε. Α, sorry λέει ο πρόεδρος. Απορρίπτεται. Αφού ήταν 28-28. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Ε, κουράστηκα κι εγώ, τι να κάνω, λέει. Λοιπόν, απο, απορρίπτεται η 48. Σαράντα 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 ναι. υπέρ κατά ναι. αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 53 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Και έτσι φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ Έληξε η ψηφοφορία. Έχουμε 45 υπέρ, 12 κατά, μία εποχή. Έγινε δεκτή η γνωμοδότηση. Ευχαριστώ και συγχαίρω τον κύριο Κρεσέντσιο Ριβελίνη. Οπότε, προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, 25. Ένωση Καινοτομίας. Μεταμόρφωση της Ευρώπης για έναν κόσμο μετά την κρίση. Συγητής ο κύριος Ζωάου Φερέιρα. Και του δίνω το λόγο. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, talvez. Ορίστε, João. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα, μήπως να περιμένουμε λίγα λεπτά για να εκενωθεί η αίθουσα από όσους δεν επιθυμούν να με ακούσουν. Και όσους. Dann würde ich auch bitten, diejenigen, die nicht zuhören wollen, die... Ε, όποιος δεν θέλει να ακούσει, παρακαλώ να φύγει ησύχως για να μπορέσει ο κύριος Φερέρα να αρχίσει την ομιλία του. Κι εγώ πρέπει να φύγω, ο ίδιος. ίδιος. tak, to proszę pana Ferreira Το λόγο έχει λοιπόν ο κύριος Ferreira. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή μας αποφάσισε να κάνει αυτή τη γνωμοδότηση για τις προκλήσεις ε, της Ευρώπης μετά την κρίση. Σε ορισμένους τομείς υπήρξαν περισσότερες προσπάθειες για την τεχνολογική καινοτομία όπως στην τομέα της υγείας, της ασφαλείας των τροφίμων καλύτερη χρήση των πηγών και πόρων, δημογραφικές αλλαγές και επιπτώσεις της νέες επιδημίες, κλιματολογικές αλλαγές, συντήρηση του ποιότητα του περιβάλλοντος. Όλα αυτά είναι παραδείγματα τομέων που είναι δικαιοδοσία της Επιτροπής μας και που δείχνουν σε ποιο σημείο είναι ζωτικό να επενδύσουμε στη νέα τεχνολογία και την καινοτομία. Τέτοιες επενδύσεις στους τομείς αυτούς είναι κάτι πολύ παραπάνω από την απλή ιδέα της χρησιμοποίησης νέας τεχνολογίας. Πρόκειται για νέες υπηρεσίες, πρόκειται για ολόκληρη επένδυση που είναι πραγματική αναγκαιότητα για να ανταποκριθούμε σε μεγάλο βαθμό στα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη αλλά και η ανθρωπότητα ολόκληρη. Στη φάση λοιπόν αυτή, επειδή πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τη γνωμοδότηση αυτή, θέλω απλώς να αναφέρω μερικές ιδέες και είμαι έτοιμος να ακούσω ιδέες και άλλων συναδέλφων που ενδιαφέρονται για το θέμα. Ας πω λοιπόν δύο-τρεις ιδέες μου για την ανακοίνωση της Επιτροπής επί του θέματος πρέπει να υπάρξει συντονισμός των προσπαθειών μας για ενδυνάμωση τους και σε επίπεδο κρατών μελών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα απορριθμιστούν οι προσπάθειες που γίνονται περιφερειακά Απλώς θα υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμό των επενδύσεων για να υπάρξει μια ανάπτυξη πιο σταθερή στην έρευνα σε όλες τις χώρες. Αυτό είναι απαράβατος όρος για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη καθώς και κοινωνική και περιφερειακή και όλα αυτά με βιωσιμότητα και συνεχή. Η μία περιφερειακή στρατηγική ανάπτυξης είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για να υπάρξουν επιπτώσεις θετικές στη προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση των του βιωτικού επίπεδου των πληθυσμών που ζουν στις περιφέρειες, για να περιοριστώ σε αυτά που είναι δική μας δικαιοδοσία. Τέτοιου είδους καινοτομία θα ήταν το βασικό στοιχείο που της δημόσιας πολιτικής, για τα ύδατα, για την παιδεία, για ένα σωρό πράγματα. Και πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια συνδυασμού. Όχι μόνο στο δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες και στην κοινωνική οικονομία. Υπάρχουν διάφορα συστήματα συντονισμού των προσπαθειών για καλύτερο συντονισμό της επιστημονικής έρευνας, παραδείγματο χάρη, αλλά αυτό δεν μπορεί να διαχωρίζεται από την παιδεία σε όλα τα κράτη-μέλη, όποιο και να είναι το τωρινό της επίπεδο και χωρίς καμία άνηση μεταχείριση από το κατώτερο μέχρι το ανώτατο επίπεδο με ιδιαίτερη έμφαση στην επιστήμη, το περιβάλλον και την υγεία. Πολλοί από αυτούς τους τομείς σήμερα έχουν τύχει επί σειρά ετών από πολύ, χαμηλές, πολύ χαμηλών επενδύσεων και έτσι δεν υπάρχει ο αριθμός που απαιτείται ειδικευμένου προσωπικού ερευνητών και ερευνητριών και έτσι υπάρχουν σήμερα φραγμοί σοβαρή φραγμή στην ενδυνάμωση των προσπαθειών που πρέπει να γίνουν για τη χρησιμοποίηση της των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας. Σας ευχαριστώ και αναμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στο Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ γενικά με την πρόταση αυτή. Όλα τα θέματα τα οποία τέθηκαν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Θα ήθελα να υπογραμμίσω όμως εδώ μια γενικότερη αντίφαση. Από τη μία βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με θέματα τα οποία έχουν αρκετά μεγάλη σημασία στο επίπεδο της Ένωσης θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με κοινά μέσα, κοινοτικά μέσα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταλήξουμε στο να κατανοήσουμε σωστά πώς, ποια είναι μάλλον η κλίμακα η κατάλληλη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και έτσι να προχωρήσουμε στις απαραίτητες πρόνοιες οι οποίες να βρίσκονται θα έλεγα στο επίπεδο της ανάγκης το οποίο αντιμετωπίζει η Ένωση. Αυτό νομίζω είναι το βασικό γιατί αλλιώς έχουμε να κάνουμε με μια προβληματική η οποία στην ουσία πολυδιασπάται στα κράτη-μέλη και δεν υπάρχει καμία συμφωνία για την κατάληξη σε ορισμένες πολιτικές οι οποίες να βρίσκουν λύσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες τις οποίες πρέπει να έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο οικονομικό. Δεν θα πρέπει να προωθούμε δράσεις σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην περίπτωση κατά την οποία μάλλον οι πόροι της, τους οποίους έχει στη διάθεσή της η Ένεση δεν είναι ανάλογοι με την σημασία και την προσπάθεια που πρέπει να γίνει. Συνεπώς, το ότι εμείς προχωράμε με ένα προϋπολογισμό της Ένωσης, ο οποίος είναι ένα προκαθορισμένο ποσό και ένα προκαθορισμένο ποσοστό του ΑΕΠ είναι κάτι το οποίο δεν θα μας βοηθήσει να λύσουμε τα προβλήματα. Γιατί κάτω από τη συγκεκριμένη προϋπόθεση δημιουργείται η εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σημασία και η παρέμβασή της και το βάρος της θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Το θέμα είναι λοιπόν να αλλάξουμε τη λογική με την οποία διαμορφώνεται ο προϋπολογισμός της Ένωσης και να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πόρους οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία η Ένωση καλείται έτσι και αλλιώ να βρει μπροστά τη. Να πω επίσης ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο πράγματι κρίσης και αντικειμενικά θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες εξοικονόμησης. Ένας λόγος παραπάνω να αναζητήσουμε εναλλακτικού πόρους, επιπλέον πόρους όπως αυτοί ε, που θα προέλθουν από την προσπάθεια που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα ευρωομόλογα. Εάν δεν υπάρξει ανάπτυξη οικονομική θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξουν ε, ε, επενδύσεις. Λοιπόν, κατά τα άλλα, όπως είπα, συμφωνώ με τις προτάσεις, αλλά θα πρέπει να βρούμε την αποφασιστικότητα που μας λείπει σαν κοινοβούλιο και να πούμε ότι αν οι προσπάθειες αυτές είναι οι ευρωπαϊκές προσπάθειες, τότε εξ αρχής η Ένωση θα πρέπει να έχει τα μέσα για να πετύχει. Ευχαριστώ. Η κυρία Μέρκες και μετά ο κύριος Αϊκάουτ. Ευχαριστώ. Όπως είπατε, λέει η κυρία Βίλμοτ, καινοτομίες, οι καινοτομίες ε, θα κατευθύνουν το καινούριο μας πρόγραμμα. Και είναι και πολύ σημαντικές οι καινοτομίες για την οικονομία μας. Βασικά για την απασχόληση. Πότε, πότε θα αρχίσει να λειτουργεί ε, το πρόγραμμα καινοτομιών. Όχι μόνο συνεργασία, αλλά και συγκεκριμένες δράσεις, αυτά που θέλουμε να επιτύχουμε. Διατομεακά δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμός όλων των τομέων στην, στις κοινωνίες μας, αλλά και ενδοκοινοβουλευτικά, ένα συντονισμός μεταξύ όλων των επιτροπών, όχι μόνο στην Επιτροπή Ίντρα, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, ΑΦΕΤ για να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια σωστή αντίδραση μέσα ε, στην Επιτροπή ε, και για να μπορέσουμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτά που θέλουμε να καταφέρουμε. Συνέχεια αναφέρουμε προκλήσεις, προκλήσεις της κοινωνίας, μεγάλες προκλήσεις. Δεν πρέπει όμως να έχουμε υπερβολικά πολλές προκλήσεις. Ας συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στον τομέα της ενέργειας, στο διοξίδιο του άνθρακα, στην σωστή απόδοση και χρήση των πόρων. Όλα αυτά πρέπει να τα ενισχύσουμε για να ξεφύγουμε, για να βγούμε από την κρίση. και επίσης βεβαίως να προσέξουμε και τον σωστό τρόπο ζωής μας, την τρίτη ηλικία, τις ποδομές κλπ. Σορία λοιπόν μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων. Πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ουσιαστικά. Θα πρέπει να αποφύγουμε τη διάσπαση αυτών των μεγάλων προκλήσεων σε πολλαπλές πτυχές Συνήθως έχουμε υπερβολική, έχουμε πλεόνασμα στόχων, υποστόχων, παραπλεύρων, δευτερεύοντων στόχων κλπ. και χάνουμε το μύτο της Αριάδνης. Η πολιτική μας θα πρέπει ίσως να καθοδηγείται από τις, τα ερευνητικά επιτεύγματα ε, ή θα πρέπει ε, να βασιστεί σε κάποια καινούργια ανακάλυψη ή σε κάποια καινοτομία ε, όπως πριν από χρόνια έγινε ας πούμε το Amazon. Mm. Θα πρέπει λοιπόν, ε, ωραίο είναι να μιλάμε για καινοτομίες αλλά θα πρέπει να έχουμε και τα κατάλληλα μέσα που θα προωθούν τις καινοτομίες, ε, που θα βοηθήσουν τις κοινωνικές προκλήσεις. Επίσης αυτές οι κοινοπραξίες μεταξύ ιδιωτικού και φορέα και επιστημονικών ιδρυμάτων. Spontaneous inventions that have not found Μπορεί να βοηθήσει κάποια καινούρια ανακάλυψη, κάποια καινούρια καινοτομία. Όταν μιλάμε για καινοτομίες, ναι, Μπορεί να είναι μια υπηρεσία, δεν χρειάζεται πάντα να είναι προϊόν. Μπορεί να είναι ένα κοινωνικό κίνημα όπως το Facebook ή μπορεί να είναι μια αλλαγή συμπεριφοράς. service We want Και θέλουμε να επιτύχουμε αλλαγή συμπεριφοράς. Και γι' αυτό θα πρέπει να ε, βάλουμε τον πολίτη σε πρώτη προτεραιότητα και σε όλες αυτές τις τέσσερις κατηγορίες καινοτομιών. Όπως ανέφερε και ο συνάδελφος Πρόντι, ο προϋπολογισμός μας, τα δημοσιονομικά μας μέσα πρέπει να ενισχύσουν τις ε, εταιρείες και τα ερευνητικά κέντρα που μπορούν να δημιουργήσουν αυτές τις καινοτομίες. Ε, πρέπει να δώσουμε ενισχύσεις σε αυτούς τους καινοτομικούς φορείς. Και επίσης να μειώσουμε το διοικητικό άχθος. άχθος αν καταφέρουμε να συνδυάσουμε ε, τη σωστή εστίαση με τους σωστούς οικονομικούς πόρους, τότε δεν θα χάσουμε τη μάχη με τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Κίνα. Χώρες οι οποίες είναι εξαιρετικά ικανές να προωθήσουν τα προϊόντα τους στις αγορές. Λοιπόν, εστίαση και οικονομική ενίσχυση για καινοτομίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μέρκες. Κύριο Σέκχουτ έχει το λόγο. Πράγματι η έκκληση για την καινοτομία είναι κρίσιμη. Καιρός είναι πλέον να προσπαθήσουμε να φανούμε κάπως πιο συγκεκριμένοι. Τα θέματα αυτά τα συζητάμε εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες. Αλλά οι δαπάνες οι ευρωπαϊκές για την καινοτομία σε σχέση με την Ιαπωνία και τη ΣΥΠΑ, η απόσταση μας με αυτούς αυξάνεται συνεχώς. Συνεπώς το πρόβλημά μας είναι σοβαρό. Πρέπει να αλλάξει η κατάσταση, πρέπει να αυξήσουμε τις διαθέσιμες πιστώσεις. Αν δούμε τους στόχους της στρατηγικής για το 2020, Μιλάμε για καινοτομία, έξυπνη ανάπτυξη, ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς μέσω των καινοτομιών. Οπότε πρέπει να έχουμε χρήματα για να τα πετύχουμε όλα αυτά. Αν δει κανείς τα θέματα αυτά περιβαλλοντικά, μια και είμαστε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και αν δούμε τα λεγόμενα flagship, της ε, ε, ναυαρχίδες αυτές σε συγκεκριμένου τομείς, ε, δεν υπάρχει γενικότερα μια συγκεκριμένη δυνατότητα. Πρέπει τουλάχιστον αυτές τις συγκεκριμένες flagships να τις χρηματοδοτήσουμε σωστά για να λειτουργήσουν σαν κινητήρια δύναμη και ε, για τους υπόλοιπους. Πρέπει λοιπόν και συμφωνώ εδώ με την εισηγήτρια να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένες προκλήσεις. Η μία είναι η γύρανση του πληθυσμού και η άλλη το πώς θα διαχειριστούμε τους διαθέσιμους πόρους. Αν δει αυτή τη στιγμή κανείς το flagship της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καινοτομία, επιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον τομέα των γερατιών με υγεία της ε, νομίζω ότι και αυτή η εταιρική σχέση η καινοτομική θα πρέπει να προωθηθεί. Ε, υπάρχουν επίσης και κάποιες άλλες προσπάθειες για τις έξυπνες μετακινήσεις, τις έξυπνες πόλεις, την αηφορία στις προμήθειες, Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με περισσότερες πιστώσεις γιατί σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν την επίτευξη των στόχων του 2020. Δεν ξεχνάμε την υγεία της τρίτης ηλικίας αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε και όλα τα θέματα αυτά. Είναι κοινωνικά προβλήματα πάρα πολύ σημαντικά. Δεν θα πρέπει να ξοδεύουμε τα χρήματά μας σε βαθμό που να μην είναι αποτελεσματικά και να μην μένουμε όσο και όσο περισσότερο περνάει ο χρόνος πίσω από τη ΣΥΠΑ, την Ιαπωνία και την Κίνα. Ευχαριστώ. Πιετικά είναι, έχει ναι, το λόγο. Ευχαριστώ. Συγχαίρω τον εισηγητή και τονίζω δύο θέματα. Πρώτον, όταν αρχίσαμε να χειριζόμαστε αυτό το θέμα, δηλαδή την υγιή γύρανση, θέλαμε να δούμε πρώτα τι αποτελέσματα θα υπήρχαν στα κράτη-μέλη ως προς την πρωτοβουλία αυτή της υγιούς γύρανσης τρία, πέντε ή ακόμη και έξι χρόνια πριν αρχίζαμε την εφαρμογή των προτάσεων to start uh, working with the resource. και να δούμε τι πόρους μπορούσαμε να κατανείμουμε. Από ό,τι κατάλαβα λοιπόν, χρειάζεται καλύτερο συντονισμός και χρήση της συνεργασίας αυτής με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με όλους τους τομείς που θέλουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που υπάρχουν για βελτίωση όλων των βιώσιμων επιχειρήσεων που δεν εκπέμπουν διοξίδιο του άνθρακος κλπ. Και με αυτό πρέπει να συνδυάσουμε και τη λύση άλλων προβλημάτων, την οποία δεν έχει κανείς από εμάς βέβαια. Η καλύτερη χρήση των πόρων είναι μία από τις σοβαρότερες ναυαρχίδες που έχουμε ποτέ φανταστεί. Και έπειτα το πρόβλημα της Ευρώπης είναι πώς θα βοηθήσει τις καινοτόμες επιχειρήσεις που αρχίζουν τη ζωή τους. Ιδίως αν είναι μικρομεσαίες οι επιχειρήσεις αυτές. Πρέπει λοιπόν να βέλτιώσουμε τη χρήση των παρακινδυνευμένων κεφαλαίων ώστε να γίνει καλύτερη χρήση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και στον τομέα αυτό και ελπίζω να το προσθέσετε αυτό στην έκθεση. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Τροπολογίες, ε, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 18 Φεβρουαρίου, ώρα 12. Επόμενο σημείο, 26. Πράσινη βίβλος της Επιτροπής. Προστασία των δασών και σχετική πληροφόρηση. Προετοιμασία των δασών εν ώψη της κλιματικής αλλαγής. Κρήτον Αρσένης. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τα δάση τα οποία καλύπτουν 42% του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλουν 10% στο βιομηχανικό ΑΕΠ, 10% των ετησίων εκπομπών, δημιουργούν 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και προστατεύουν το έδαφος, από τη διάβρωση, τις πλημμύρες κλπ. Η πρώτη έκθεση του Κοινοβουλίου ήταν η έκθεση Τόμας το 1997 για την δασοκομεία και τη στρατηγική της δασοκομείας. 40 σελίδες είχε η έκθεση αυτή που ζητούσε την ανάπτυξη και υποστήριξη συντήρηση των δασών. Σήμερα έχουμε πολλές πολιτικές και οικονομικά μέσα που αφορούν την δασοκομεία. Περιβαλλοντική νομοθεσία, βιοπικιλότητα, ε, νομοθεσία ενεργειακή, τα, ταμείο συναχής, πολιτική προστασία. Ένα μεγάλο πλαίσιο μέτρων δηλαδή. Όταν συζητήσουμε ε, την ποιότητα της ατμόσφαιρας Ζητήσαμε την προστασία των δασών και σε, πάνω σε αυτό το θέμα βασίζεται, βασίζονται και πολλές περιβαλλοντικές δράσεις. Η πρώτη στρατηγική προστασία δασών υιοθετήθηκε το 1998 και 8 χρόνια αργότερα το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δασοπονίας το οποίο είχε τέσσερις βασικούς στίχους. Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, ε, βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος, βελτίωση και προστασία ποιότητας ζωής και ενίσχυση επικοινωνίας, πληροφόρησης. Από τους τέσσερις στόχους, η αξιολόγηση του προγράμματος δράσης δασοπονίας δείχνει ότι ενισχύθηκε η ανταγωνιστικότητα, βελτιώθηκε λίγο η πληροφόρηση, αλλά πολύ λίγη πρόοδος έγινε στην ε, προστασία και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οπότε, ένα πράγμα που ζητήσαμε να περιληφθεί στην πράσινη βίβλο ήταν η προστασία περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Και η Πράσινη Βίβλος επίσης ζητήσαμε από την Πράσινη Βίβλο να μας βοηθήσει να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή. Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες δασοκομείας ε, λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Όμως η κλιματική αλλαγή παρουσίασε νέες απειλές από αυτές ε, και εάν κανείς μελετήσει τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Δασοκομικού Ινστιτούτου θα δείτε ότι πολλές αρνητικές επιπτώσεις ε, παρουσιάζονται στον γεωργικό τομέα. Ε, ε, αλλαγή του κλίματος, πλημμύρες, πυρκαγιές και οι επιπτώσεις αυτών των φαινομένων είναι σωρευτικές διότι οδηγούν και στην ε, ε, ε, υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους αλλά και στη μείωση των δασών. Οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα φαινόμενα που υπάρχουν, που, που σημειώνονται. Οι, τα δάση αναπτύσσονται σε, σε πέντε κλιματικές ζώνες. Η Μεσόγειος, η αλπική περιοχή, τα Καρπάσια, τα οράλια και αυτές οι πέντε δασικές περιοχές, σε αυτές πρέπει να εφαρμόσουμε τα 14 κριτήρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Και πρέπει να εφαρμοστούν κοινά μέτρα σε αυτές τις πέντε δασικές ζώνες. Ανανέωση λοιπόν των δασών, αυτό είναι ένα μέτρο που πρέπει να ενισχύσουμε. Αναμόρφωση, ανανέωση, αναδάσωση, ε, χρησιμοποίηση νέων υλικών, ε, σωστή διαχείριση των δασών, κοπή κλάδων, αρέωση, ε, νέες φυτεύσεις νέοι τρόποι διαχείρισης των δασών, και λοιπά. Για την προστασία των δασών ε, πρέπει να ενισχύσουμε την φύτευση διαφορετικών ειδών δέντρων ώστε να υπάρχει μια ποικιλία και ε, ε, δεδομένου ότι έχουμε αυτές τις εκθέσεις και τις γνωμοδοτήσεις της Ήτρε και του Σάγκρη και μετά από όλες τις εργασίες που έχει διοργανώσει το Κοινοβούλιο και ευχαριστώ ιδιαίτερα τη γραμματεία της Επιτροπής μας εδώ και τους συναδέλφους και επίσης ε, όλους τους, τους ενδιαφερόμενους με τους οποίους είχα τη δυνατότητα να συνεργαστώ για να συντάξω τη γνωμοδότησή μου. Τους ευχαριστώ λοιπόν όλους. Η βασική αντίδραση, πρέπει να απαντήσουμε σε αυτές τις προκλήσεις με τρεις ε, νομοθετικές προτάσεις. Η μία πρόταση είναι καινούρια. Και λέει το εξής. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα νέο πλαίσιο προσαρμογής δασών και αυτό να αποτελεί την κοινή βάση προστασίας του δασοκομικού πλούτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παρουσιάζει μέτρα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και συντήρηση των δασών, κατευθυντήριες γραμμές για μία αριφόρο ανάπτυξη δασών και αυτό λοιπόν το καινούργιο πλαίσιο θα πρέπει να έχει μία νομοθετική ισχύ ε, και να εφαρμοστεί σε όλο το, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να εκπονηθούν υποχρεωτικές εθνικές πολιτικές για την δασοκομική πολιτική δύο, άλλα, δύο άλλες νομοθετικές προτάσεις για τις πυρκαγιές δασών και για την πληροφόρηση, ενημέρωση, έχουν εκπνεύσει. Προτείνω λοιπόν μία, ένα τρίτο νομοθετικό πλαίσιο για, για τις πυρκαγιές, πρόληψη, καταπολέμηση κλπ. και ενημέρωση πολιτών. Η ύπεθρος, η, η ύπεθρος, όπως σας είπα, η ευρωπαϊκή ύπεθρος καλύπτεται κατά 42% από δάση. Και πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε τρόπους ε, χρηματοδότησης στον πρώτο πυλώνα, ιδιαίτερα να ενισχύσουμε μονάδες παραγωγών, όπως προτείνει και η Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων, η Αγκρή, αλλά και το, τους δημόσιους ε, τομείς ε, για να μπορέσουν να προστατεύσουν τα δάση από τις κλιματικές αλλαγές. Ε, Επίση, πρέπει να βρούμε τα απαραίτητα κονδύλια για την εξασφάλιση της βιοπικιλότητας και των ερευνών των οι μελέτες, οι έρευνες που πρέπει να γίνονται στα δάση πρέπει να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένε δασικές ζώνες, να, να είναι δηλαδή επικεντρωμένες στο συγκεκριμένο έδαφος και στις συνθήκες που επικρατούν σε αυτές τις δασικές ζώνες. Και τέλος, όσον αφορά τώρα το ζήτημα των εκπομπών, η πρόταση που σας υποβάλλω είναι να μην προτείνουμε στο ETS αυτά τα στοιχεία, διότι το ITS ε, εργάζεται σε αιτήσια βάση, ενώ το LUTS ε, χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσει αυτά τα αποτελέσματα και είναι πολύ δύσκολο ε, για να κρίνουμε τις βιομηχανικές εκπομπές, να, να τεμαχίσουμε ένα δάσος σε συγκεκριμένες ιδιοκτησίες. Πρέπει να λάβουμε, να ξανασκεφτούμε την ουδετερότητα άνθρακα σε σχέση με τη, με τη βιομάζα. Εάν θέλουμε να έχουμε σωστές, σωστά μετρήσιμα στοιχεία της εξοικονόμησης εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, πρέπει να έχουμε και νομοθετικά μέτρα ε, υποχρεωτικά για τη βιομάζα. Και αυτά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα έχουμε. Αλλά πρέπει να έχουμε σαφείς ορισμούς των δασών, δεδομένου ότι υπάρχουν διάφορες μορφές δασών, νέες φυτίες, παραδείγματος χάρη, παλαιά δάση, ε, πρέπει να έχουμε ξεκάθαρους ορισμούς. Ε, σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να καταλήξουμε σε μια πολύ σωστή, πολύ καλή γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο εισηγητή. Έχουν ζητήσει αρκετοί συνάδελφοι το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα πρέπει να είμαι ιδιαίτερα σύντομη γιατί έχει περάσει η ώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί μπόρεσε να αντιμετωπίσει αυτό το πάρα πολύ περίπλοκο και ενδιαφέρον θέμα. Είναι περίπλοκο για πολλούς λόγους το θέμα του. Από τη μία είναι σαφές ότι έχουμε ανάγκη τέτοιου είδους εκθέσεις γιατί θα τις χαρακτήριζα υποδειγματικές αφορούν την κατάσταση των δασών στην Ευρώπη και την προετοιμασία τους στις κλιματολογικές αλλαγές. Διαπιστώνουμε ότι σήμερα έχουμε αρκετά στοιχεία στη διάθεσή μας και μπορούμε να υπολογίσουμε τις συνθήκες οι οποίες θα διασφαλίσουν την προσαρμογή στις κλιματολογικές αλλαγές και στη βιοπικιλότητα. Τα αποθέματα δασών, σε εισαγωγικά τα αποθέματα στην Ευρώπη, πιέζονται γιατί χρησιμοποιούνται και για την παραγωγή βιομάζας. Το θέμα είναι ε, να δούμε τι ποσότητα βιομάζας προέρχεται από την εκμετάλλευση την δασική θα πρέπει να ε, υπάρχει έλογη χρήση αυτής της δυνατότητας και να μην φτάσουμε σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα και θα καταθέσω τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί λοιπόν γιατί από τη μία θα ξοδέψουμε χρήματα για την ανανέωση των δασών και από την άλλη εμείς οι ίδιοι ξοδεύουμε τα χρήματά μας στην ουσία εξοδεύοντας τεράστιες δασικές επιφάνειες γιατί μετατρέπονται σε ε, παραγωγή βιομάζας. Σχετικά τώρα με την βιολογική ισορροπία. Νομίζω ότι αυτή είναι η προϋπόθεση εκ των ουνάνευ. Τα δάση θα πρέπει έτσι να κρατήσουν το οικονομικό και κοινωνικό τους ενδιαφέρον. Θα πρέπει να υπάρξει αηφόρος ανάπτυξη των δασών αυτών και θα πρέπει να βασιστούμε σε σωστούς τρόπους διαχείρισης τεχνικής των δασών. Η εκμετάλλευση των δασών υπάρχει και θα υπάρχει. Πρέπει λοιπόν να επιστήσουμε την προσοχή όλων των εμπλεκομένων στο ότι επικρατούν μερικές φορές διαφορετικοί ορισμοί και διαφορετικές ε, ιδέες για το τι είναι δάσος, για το τι είναι δασική έκταση είναι απαραίτητο να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στους ορισμούς τους οποίους χρησιμοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων ή ίσως και σε κάποιους άλλους ορισμούς οι οποίοι ε, είναι καρπό σοβαρή επεξεργασίας, γιατί αλλιώς φοβάμαι θα δημιουργηθούν πολλές συγχύσεις και δεν θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα εδάφια αυτά αποτελεσματικά. Υποστηρίζω λοιπόν την πρόταση του εισηγητή έτσι ώστε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστούν καλύτερα ε, σε επίπεδο ε, δασικών εκτάσεων και με τις δασικές υπηρεσίες. Όλα αυτά εντάσσονται στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος για την εκμετάλλευση και την πρόοδο της υπαίθρου. Εδώ έρχονται και οι κοινωνικές πλευρές. με την άποψη του εισηγητή λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας κάνει μια πρόταση και για το θέμα πλέον της πρόληψης των πυρκαγιών στα δάση. Γνωρίζουμε τι τεράστιες επιφάνειες έχουμε χάσει μέχρι τώρα λόγω άγνοιας, ίσως και λόγω προκλήσεων και πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σοβαρό τρόπο το θέμα των πυρκαγιών και της πρόληψης των πυρκαγιών. Εδώ απαιτείται να υπάρξει και οικονομική στήριξη και για τη σωστή ενημέρωση αλλά και για τα συστήματα προειδοποίησης κάτω από πολλές μορφές. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ο έλεγχος της λειτουργίας των δασών και ο ρόλος τους στα πλαίσια των κλιματολογικών αλλαγών. Ευχαριστώ κύριε Χούμναρ. Όκεν. Και μετά Κάλαχαν. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον κύριο Αρσένη για τη δουλειά του επ' αυτού του ιδιαίτερα σημαντικού θέματος. Τα δάση φυσικά είναι ένα κλειδί της γεωγραφίας της Ευρώπης. Δεν είναι σημαντικά μόνο από περιβαλλοντολικής απόψεως, αλλά προσφέρουν πάρα πολλά ωφέλη και υπηρεσίες από τις οποίες υποφελούμαστε πολύ όπως είπε δικαίως, δημιουργούν θέσεις εργασίας και πρώτες ύλες για την βιομηχανία και για ανανεώσιμες πηγές ενεργείας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που τόνισε τη σημασία των πολλών, ε, τη μεγάλη σημασία που έχουν τα δάση για την απασχόληση. Επίσης, για την προστασία της βιοπικιλότητας, για τη διευθέτηση του προβλήματος της ποιότητας του εδάφους και των υδάτων. Επίσης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική κληρονομιά πολλών εθνών μας. Λόγω λοιπόν του ρόλου αυτού, καθώς και του της σημασίας που έχουν για πολλούς από τους πολίτες ακόμη και με όρους τουρισμού πρέπει να προστατευτούν. η ομάδα μου δέχεται οποιοδήποτε μέτρο προωθεί την προστασία των δασών και μεταξύ αυτών και την καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών. Δεν έχω βέβαια πλήρως πιστεί από την πρόταση του εισηγητή ότι, χρειάζεται, ότι χρειάζονται περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις από την Κομισιόν. Πρέπει πάντοτε να προσέχουμε να μην υπερχρησιμοποιούμε το νομοθετικό εργαλείο αλλά να βλέπουμε πάντοτε και πρωτίστως εάν μια ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρόσφερε τίποτε παραπάνω από αυτά που μπορεί να κάνει το, ένα κάποιο κράτος μέλος. Ο εισηγητής σημειώνει ότι διαφέρουν πολύ και οι εκτάσεις και η σημασία των δασών από χώρα σε χώρα και ακόμη δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιες επιπτώσεις θα έχει επί των δασών η κλιματολογική αλλαγή. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών, όπως λέει και ο εισηγητής, μέσω της διεύρυνσης των γνώσεων που έχουμε για τα δάση και ίσως και για το ρόλο που μπορούν να παίξουν στην καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών. Τελικά δέχομαι την έκθεση του εισηγητή και αναμένω μαζί με τις άλλες πολιτικές ομάδες να δω τι θα πούν οι συντονιστές για, με βάση όμως την αρχή της επικουρικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Όκεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω σύντομα ότι και εμείς υποστηρίζουμε πλήρως την έκθεση αυτή που χρειαζόταν πράγματι διότι τα δάση παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, πολλές φορές παραγνωρίζονται. Όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να παραμείνουν εν ζωή τα δάση. Και γι' αυτό εμείς υποστηρίζουμε και τις συστάσεις του εισηγητή. Αυτό ήθελα μόνο να πω και τον ευχαριστώ εκ νέου. Ευχαριστώ κυρία Άουκεν η κυρία Ντεμπρά και μετά η κυρία Κατρίν Σολή. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κρήτον Αρσένη για το πάρα πολύ χρήσιμο σχέδιο γνωμοδότησης που καλύπτει πάρα πολλά ζητήματα που συζητάμε. Όλοι αναγνωρίζουμε την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική σημασία των δασών μας και ε, βεβαίως Επίσης ε, αναγνωρίζουμε ότι η δασοκομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξαιρετικά περίπλοκη και επίσης ότι πάρα πολλές άλλες πολιτικές επηρεάζουν τα δάση και αντίστροφα και τα δάση, η δασοκομική πολιτική μπορεί να έχει επίδραση στον τουρισμό, σε κοινωνικές ε, αλλαγές, σε οικονομικές ε, σε οικονομικά ζητήματα κλπ. Άκουσα το Κρήτονα να μιλάει με πολύ ενθουσιασμό για τα επιτεύγματα του, της Ναγκόγια και ίσως θα έπρεπε στις διάφορες παύλες να περιληφθεί και η Ναγκόγια, τα συμπεράσματα. Επίσης, αναφέρθηκε στα οικοσυστήματα, αναφέρεται στην έκθεσή του στα οικοσυστήματα. Ε, εγώ πιστεύω ότι τα δασικά οικοσυστήματα πρέπει οπωσδήποτε να ισχυθούν για να προστατευτούν τα δάση από τη διάβρωση του εδάφους, ε, τις κλιματικές αλλαγές κλπ. Ίσως λοιπόν καλό θα ήταν να γίνει μία αναφορά στο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Θα μπορούσε αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο να χρησιμοποιηθεί για την βιωσιμότητα των και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων. Ε, Δύο-τρεις άλλες παρατηρήσεις. Ε, έχει εξαιρετική σημασία να αναγνωρίσουμε τους τέσσερις στόχους που πρέπει να εφαρμόσουμε, αλλά πέραν από αυτούς χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους στόχους και μέτρα για το περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής Επίσης, η αρχή της επικουρικότητας στην παράγραφο 1 αναφέρεται σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, λέει παράγραφος 1. Μήπως θα μπορούσε ο Κρήτον λίγο να μας εξηγήσει το, το 14 το 14 που αφορά την προστασία των δασών από πυρκαγιές. Πώς, μπορεί, πώς θα εφαρμόζεται ή πώς επηρεάζεται η αρχή της επικουρικότητας στα πλαίσια της ε, πολιτικής προστασίας. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να ευθυγραμμίσουμε ε, περισσότερο ε, την ε, πολιτική προστασία περιλαμβάνοντας και την αρχή της επικουρικότητας. Επίσης το γενετικό υλικό, πολύ σημαντικό. Έχει οικονομική πτυχή, σαφώς, αλλά μην κοιτάμε μόνο τα οικονομικά θέματα και την αντιγωνιστικότητα, αλλά και την προσαρμοστική ικανότητα του δάσους. Γι' αυτό το γενετικό υλικό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Συμφωνώ ε, σαφώς ότι δεν πρέπει να έχουμε το LULUCF στο ICF και ε, συμφωνώ γενικά και σε άλλα ζητήματα της έκθεσης. Τα βασικά είναι πρώτον, ναγκόγια στις Παύλες, ενίσχυση της δασοκομείας, του ρόλου της δασοκομείας, έρευνα και τεχνολογία και συγκεκριμένη αναφορά στις νέες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολιτική προστασία. Αυτά ήταν τα τρία βασικά σημεία. Και συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι είναι μια ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο γνωμοδότησης. Ευχαριστώ την κυρία Ντεμπρά. Η κυρία Σόλη και ο τελευταίος ομιλητής ο κύριος Σπερέλο. Η κυρία Σουλή. Η έκθεση είναι πολύ πυκνή και αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον του εισηγητή για το θέμα. Τρία σχόλια τα οποία όμως δεν διαφωνούν με το κείμενο και σίγουρα θα καταθέσω και τροπολογίες. Για το σημείο 13 βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα την ιδέα της εφαρμογής ε, μια πληρωμής για την αναδάσωση αλλά πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση μεταξύ των κονοφόρων και των υπολείπων δέντρων, γιατί τα κονοφόρα δεν αλλάζουν το έδαφος τόσο πολύ όσο τα υπόλοιπα μέσα της δημιουργίας ε, εναποθέσεων στο έδαφος. Γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια διαφοροποίηση. Άλλο στοιχείο το 14 που το ανέφεραν πολύ για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Στο νότο της Γαλλίας, δυστυχώ έχει φύγει ο Φράγκο αλλά θα μπορούσε να το πει και εκείνος, έχουμε αστικές περιοχές και δασοφόρες περιοχές. Και στις ζώνες αυτές νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει εκχέρσωση για να βελτιωθεί η κατοίκηση και για να εμποδιστούν οι πυρκαγιές εκχέρσωση από ζυζάνια. Αυτό θα βελτίωνε και την οικονομία και το περιβάλλον. Στις ζώνες αυτές, όσο και αν είναι αραιοκατοικημένες, θα έπρεπε να υπάρξει αυτή η εκχέρσωση. Και τελευταίο, έχουμε τα λεγόμενα arbre remarkable, δηλαδή γίνεται προστασία ορισμένων ειδών δέντρων, συνήθως πολύ γυρεών, που έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία ή που είναι ιδιαίτερα όμορφα και τα οποία προστατεύονται. Θα μπορούσε να γίνει μια καταλογογράφηση τέτοιων δέντρων στο σύνολο της Ένωσης και στο δική μου εκλογική περιφέρεια έχουμε τρία τέτοια δέντρα που είναι καταπληκτικά. Αυτή είναι μια ιδέα που προτείνω στον εισηγητή, τον οποίο ευχαριστώ εκ Ευχαριστώ. Την κυρία Σουλή. Και εμεί στην Πολωνία έχουμε ένα τέτοιο κατάλογο ε, πολιτιστικών ε, μνημείων που, πρέπει να προστατευτούν. Ο κύριος Περέλο Ροντρίγκες παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ συμφωνώντας με τους προηγούμενους ομιλητές τον εισηγητή. θα ήθελα να επιμείνω λίγο στις συστάσεις οι οποίες γίνονται για μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα. Όταν μιλάμε για τα δάση μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις οι οποίες ε, αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο κομμάτι της, ε, του ευρωπαϊκού εδάφους, μπορεί να φτάνει το 45-48%. Και εκπλήσει το ότι δεν υπάρχει μια συνολική νομοθεσία που να καλύπτει όλες τις χώρες. Υπάρχουν διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις, διαφορετικά κριτήρια σε κάθε χώρα και υπάρχει και η αρχή της επικουρικότητας που περιπλέκει κάπως την κατάσταση. Προφανώς και υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε όπως το ζητάει και η έκθεση ότι απαιτείται να υπάρξουν κοινοί κανόνες με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας και με σεβασμό των διαφορετικών τυπολογιών των δασών. Αν χρησιμοποιούμε συστηματικά τα δύο αυτά θέματα απλά σαν άλοθη για να μην καταλήγουμε σε κοινού κανόνες τότε φοβάμαι ότι έχουμε αποτύχει. Οι κλιματολογικές αλλαγές δεν γνωρίζουν σύνορα και εμείς δεν κάνουμε τίποτα το οποίο να βελτιώνει την κατάσταση. Απαιτείται να κατανοήσουμε το τι προσφέρουν τα δάση στα πλαίσια της καταπολέμησης των συνεπειών α, της υπερθέρμανσης. Πρέπει λοιπόν κάποιες από τις τροπολογίες να βοηθήσουν έτσι ώστε το ε, κείμενο να γίνει πιο συγκεκριμένο και είναι καιρός πια να υπάρξουν κοινοί κανόνες. Τα πλαίσια πάντα βέβαια και τη σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Δύο μιλητές έχω ακόμα. Ο κύριος Πρόντι έχει το λόγο και μετά Φερέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τον συνάδελφο Κρήτον Αρσένη για την έκθεσή του. Συμφωνώ εν πολλής με αυτά τα οποία λέγει. Να μου επιτρέψετε να κάνω κάποιες μικρές παρατηρήσεις. σχετικά με τις νέες προκλήσεις τις οποίες θέτουν οι κλιματολογικές αλλαγές στο σύνολο του ευρωπαϊκού εδάφους και ιδιαίτερα στα δάση. Υπάρχει καταρχάς μία αύξηση της περίοδου ξηρασίας και αύξηση των πιθανοτήτων, των πιθανοτήτων πυρκαγιάς. Συνεπώς πρέπει να αυξηθεί η φροντίδα του δάσους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται με την βιομάζα η οποία ανακτάται από τα δάση κάτι το οποίο επηρεάζει και τη σώρευση άνθρακα στα δάση και κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει ε, σε μια μεγαλύτερη κατακράτηση άνθρακα μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη μας ότι ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές έχει πολύ μεγάλη σημασία να χειριστούμε το έδαφος με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ε, το έδαφος να κρατά το νερό όταν βρέχει με τον περισσότερο χρόνο ε, που μπορεί αυτό να γίνει, όσο περισσότερο γίνεται. Και αυτό θα βοηθήσει την ανανέωση και την ε, πλήρωση των ε, υπόγειων πόρων, υδάτινων πόρων. Λοιπόν, τα δάση όπως βλέπουμε παίζουν σημαντικό ρόλο και στον κύκλο αναπαραγωγής και αναπλήρωσης του ύδατος. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από ένα σύστημα παρακολούθησης ε, πάρα πολύ λεπτόμερες. Έχουμε ήδη το πρόγραμμα δορυφορικής παρακολούθησης για την ασφάλεια και το περιβάλλον. Είναι κάτι το οποίο νομίζω μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις απειλές οι οποίες αυτή τη στιγμή, τις οποίες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τα δάση. Είναι απαραίτητο να μπορούμε να τα παρακολουθούμε από κοντά, γιατί τότε μόνο θα μπορέσουμε ποσοτικά να προσμετρήσουμε το στρες το οποίο υφίστανται οι δασικές εκτάσεις και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσουμε κοινοτικά και όχι σε εθνικό μεμονωμένο επίπεδο. Το ευχαριστώ κύριε Πρόντι και ο τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Φεραίρα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο, τον Αρσένη για την ε, παρουσίασή του, την εισήγησή του και τις διάφορες προτάσεις του. Ε, θετικές προτάσεις, ιδίως ε, στην αρχή της επικουρικότητας. Και επίσης υπάρχει το θέμα της απαραίτητης διάκρισης η οποία θα πρέπει να γίνει ανάμεσα στις διαφορετικές τυπολογίες που χαρακτηρίζουν τα δάση. Αυτόχτονα δάση κτλ. Ε, δάση μονοκαλλιέργειας, διαχειριζόμενα δάση κτλ. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες και ε, θα ήθελα να τονίσω δύο ίσως επιπλέον στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα για τον εισηγητή. Από τη μία Υπάρχει η κατάσταση των δασών σε επίπεδο φυτοϊγιεινής. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία απειλούν ορισμένα είδη ε, φυτών και ε, προβλήματα τα οποία προέρχονται από, ορισμένα, ε, από ορισμένες κατηγορίες εισβολέων, φυτοεισβολέων θα τους έλεγα. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε ακριβώς με σωστό έλεγχο. Ένα άλλο θέμα το οποίο δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα είναι η πρόληψη των φυσικών καταστροφών. Σας θυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε υιοθετήσει μια έκθεση το 2010 για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών. Είχαμε κάνει μια ολόκληρη σειρά από προτάσεις οι οποίες καλύπτουν και τα δάση. Πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει συνέχεια σε αυτές τις συστάσεις. Είναι λοιπόν απαραίτητο να ζητήσουμε από τον εισηγητή να επανέλθει σε αυτές τις προτάσεις που είχαμε κάνει. Θυμίζω ότι είχαν προταθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι οποίες δεν έχουν ακόμα ληφθεί. Είναι απαραίτητο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην αγνοήσει αυτά τα οποία είχαμε προτείνει και να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της. Επίσης θα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά το θέμα της αποκατάστασης των δασικών περιοχών που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές. Αυτό ισχύει για περιοχές όπως η Μεσογειακή Ευρώπη, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία κτλ. Πρέπει να προωθούμε ε, αυτόχτονα ήδη για την αντικατάσταση των ζημιών στα δάση βέβαια. Ευχαριστώ τον ε, κύριο Φερέιρα Νομίζω ότι η προθεσμία κατάθεσης των απολογιών είναι η 9η Φεβρουαρίου 2011, τη 12η μεσημβρινή. Το 27 αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 97-68 όσον αφορά τις διατάξεις τους κινητήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος. Εισηγείται η κυρία Πιατεκάινεν. Έχετε το λόγο. Uh, ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω την υπομονή των συναδέλφων, δεδομένου ότι η ώρα είναι προχωρημένη, να σας εξηγήσω λίγο περί τίνος πρόκειται. Και τι προτείνω. Καταρχάς, η οδηγία για τους κινητήρες, μη οδικούς κινητήρες, περιλαμβάνει και καλύπτει πολλούς κινητήρες που χρησιμοποιούνται στον οικοδομικό τομέα, στη δασοπονία, σε κινητήριες μηχανές, στην οδοπία και αυτή η οδηγία του 2004 είχε ως σκοπό να εισαγάγει νέα όρια εκπομπών και ένα σύστημα ευέλικτο που θα επιτρέπει στους κατασκευαστές να διαθέσουν στην αγορά έναν περιορισμένο αριθμό μηχανημάτων τύπου 3α, παλαιότερου τύπου δηλαδή. Η ευελιξία τώρα είναι ή 20% του, του, του όγκου παραγωγής των κατασκευαστών ή ένα συγκεκριμένο ποσοστό για συγκεκριμένο μηχάνημα. Συγκεκριμένο κινητήρα μάλλον. Γιατί οι κατασκευαστές παράγουν έναν περισμένο αριθμό κινητήρων γιατί πρόκειται για μεγάλα μηχανήματα και αυτό που προτείνω εγώ uh, uh, uh, και που μπορείτε να διαβάσετε στην γνωμοδότησή μου είναι το εξής. Η Κομισιόν θέλει να αυξήσει το 20% ευελιξίας σε 50% και να τροποποιήσει τους σταθερούς ε, αριθμούς, τα σταθερά στοιχεία αντίστοιχα. Για ορισμένους λόγους εγώ δεν συμφωνώ με την αύξηση του στοιχείου ευελιξίας από 20% σε 50% αλλά συμφωνώ μόνο με την αύξηση συγκεκριμένων αριθμητικών στοιχείων. Εάν έχετε την πρόταση στα χέρια σας, μπορείτε να δείτε στον πρώτο πίνακα τον ε, αριθμό των κινητήρων, την κατηγορία στην οποία ανήκουν με το 20% και στον δεύτερο πίνακα το, στο 1.2.2 οι νέες προτάσεις με τα στοιχεία της Κομισιόν. Ε, βλέπετε λοιπόν συγκρίνοντας τον πίνακα και τις προτάσεις Κομισιόν υπάρχει μία αύξηση ανά κατηγορία, ανά κατασκευαστή, την οποία δέχομαι. Επίσης προτείνω να αποκλειστεί ο κατασκευαστικός, ο οικοδομικός τομέας από, αυτό, από αυτή την ευελιξία διότι σε αυτόν τον τομέα παρουσιάζονται δυσκολίες ε, όσον αφορά τον σαφή ορισμό των κινητήρων για την εξασφάλιση της μεταχείρισης. Να, να, να, να είναι απ' να ε, εξαιρεθεί ο κατασκευαστικός τομέας. Προτείνει λοιπόν η Κομισιόν για τις ε, μηχανές των τρένων 50% ευελιξία. Εγώ προτείνω να μην συμπεριλάβουμε στο σύστημα ευελιξίας ε, τους ιδρομικούς σειρμούς και για τις, ε, τους ε, κινητήρες για τους σειρμούς φορτίων προτείνω ε, ακόμα ένα μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που προτείνει η Κομισιόν, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένε ε, καταστάσεις στο Ενωμένο Βασίλειο. Εδώ πρέπει να προσαρμόσουμε ε, την σύνταξη του κειμένου για να προσαρμοστεί στην κοινωτική νομοθεσία. Και αναμένω με ανυπομονησία τις προτάσεις σας. Σύμφωνα με την ανάλυση της Κομισιόν, Οι περισσότεροι από τους 1.500 κατασκευαστές μη οδικών κινητήρων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ε, αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως πάντα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες από ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις ιδίως όσον αφορά στην προσαρμογή συμβατότητας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να υπάρχει περισσότερο, περισσότερο, ένα μεγαλύτερο σύστημα ευελιξίας για, τους, για τα συγκεκριμένα, για τα οριστικά ε, στοιχεία τα οποία θα διευκολύνουν την ε, μείωση του ε, σχεδιαστικού κόστους. Τώρα, γιατί δεν συμφωνώ με την πρόταση της Κομισιόν για αύξηση από 20% σε 50% του ευέλικτου συστήματος. Ε, η Κομισιόν λέει ότι προτείνει την αύξηση του ευέλικτου στοιχείου λόγω της οικονομικής κρίσης. Πιστεύω ότι αν το δεχτούμε θα δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο διότι σε άλλες περιβαλλοντικές νομοθεσίες δεν αποδυναμώνουμε τους ισχύοντες κανόνες επειδή υπάρχει οικονομική κρίση, άρα λοιπόν γιατί να το κάνουμε εδώ. Δεύτερον, ε, οι κατασκευαστές και ο τομέας είχαν πάρα πολύ καιρό στη διάθεσή τους να προσαρμοστούν. Εάν τώρα τους παραχωρήσουμε ένα, μια μεγάλη αύξηση του ευέλικτου συστήματος, αυτό το οποίο τελικά θα, θα κάνουμε είναι να τιμωρήσουμε αυτούς που έχουν ε, σεβαστεί ε, την νομοθεσία και θα ωφελήσουμε αυτούς που δεν την έχουν σεβαστεί. Ε, δεν πρέπει λοιπόν τους αρχικούς κατασκευαστές να τους τιμωρήσουν που έχουν ήδη κάνει όλη την έρευνα και ε, την ανάπτυξη, το R&D δηλαδή, όλο το σχεδιασμό των κινητήρων σωστά ε, και συμβατά με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν πρέπει λοιπόν αυτούς να τους τιμωρήσουμε. Τρίτον, ε, όπως ξέρετε όλοι έχουμε φιλόδοξους στόχους να προχωρήσουμε προς κοινωνίες χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και βεβαίως τονίζουμε συνέχεια τις καινοτομίες με νέα νομοθετικά μέτρα κανονισμούς κλπ. Εάν λοιπόν εγκρίνουμε αυτή την αύξηση, στέλνουμε ένα εντελώς ε, λανθασμένο μήνυμα, εάν αυξήσουμε το περιθώριο ευελιξίας. Αντί να είμαστε πιο αυστηροί, είμαστε πιο ελαστικοί. Τέταρτον, στον ε, κατασκευαστικό τομέα ήδη παρουσιάζεται μία ανάκαμψη. Άρα λοιπόν τα επιχειρήματα, οι δικαιολογίες οικονομικής κρίσης δεν ευσταθούν πια τόσο πολύ. Και πέμπτον, η πέμπτη, ο πέμπτος λόγος για τον οποίο δεν συμφωνώ είναι ότι η Κομισιόν ανέμενε να κάνει την αξιολόγηση της υπάρχουσας οδηγίας και τις προτάσεις της νέας φάσης μέχρι τώρα, αλλά έχει καθυστερήσει. Θα έχουμε την αξιολόγηση και τις νέες προτάσεις φέτος. Είναι μια δυσάρεστη κατάσταση αυτή για τον τομέα και για μας. Πώς θα πάρουμε αποφάσει τώρα, εν συνεχεία θα γίνει αναθεώρηση της οδηγίας από την Κομισιόν και ίσως αναγκαστούμε να λάβουμε εντελώ διαφορετικέ και αντίθετες αποφάσεις. Είναι λοιπόν πρόωρο αυτό, όλο αυτό το θέμα. Η έκτη μου είναι περιβαλλοντική. Ο Επίτροπος Ποτότσνικ έκανε μία ανακοίνωση πριν από μερικές μέρες που είπε ότι η ατμοσφαιρική ποιότητα είναι ένας, ένα πιεστικό θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί η Κομισιόν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση για να καθιερώσουμε ε, κοινοτικά πρότυπα, ευρωπαϊκά πρότυπα για καύσιμα, για μείωση των εκπομπών από μηχανήματα, κινητήρες και οχήματα. Και ότι οι τιμές αυτές θα πρέπει να βασίζονται στους διάφορους κλάδους της βιομηχανία, των κατασκευαστικό, των μεταφορών κλπ. Και πάλι τώρα στο περιβάλλον. Η Κομισιόν λοιπόν δεν έχει λάβει υπόψη επαρκώς την ε, μακροβιότητα αυτών των κινητήρων. Και οι επιπτώσεις ε, των τοπικών εκπομπών ε, καυσαερίων είναι μεγαλύτερες από αυτά τα οποία αναφέρει. Λοιπόν, και για το κατασκευαστικό τομέα και για τον συνδρομικό τομέα τα οριστικά, οι οριστικές τιμές ε, είναι εφαρμόσιμες, είναι βιώσιμες. Ε, ο κατασκευαστικός τομέας προτείνω να εξαιρεθεί ε, και επίσης προτείνω να μην συμπεριληφθούν οι κινητήρες τρένων. ο βασικός λόγος που το προτείνει αυτό η Κομισιόν αναφέρεται στην ιδιαιτερότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και στο συνδρομικό τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αλλαγή, η τροποποίηση λέει ότι ο αριθμός των συνδρομικών και μη κινητήρων που θα πρέπει να περιληφθούν ε, πρέπει να είναι 20 maximum. Ε, και επειδή χρειάζεται ακόμα ορισμένες προσαρμογές ε, αυτής της πρότασης, εκκρεμεί το ζήτημα αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους και περιμένω με ανυπομονησία τις προτάσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ μάλιστα. Έχουμε 10 ομιλητές. Γι' αυτό σας παρακαλώ να μην μιλήσετε για πάνω από ένα λεπτό γιατί έχουμε κι άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ε, είναι. Karin Kadenbach, Elisabeth Gardini. Yeah, but it's possible that you start with the, with the shadows of the group. Because you didn't talk about the shadows of the groups. Zaczynam. Zaczynam od pana Pawła po Θα δώσετε το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές των πολιτικών ομάδων καταρχάς. Αυτό θα κάνω, είπε ο Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο καταρχάς στους συναδέλφους από τις πολιτικές ομάδες. Είναι σαφές ότι ελέγχεται ένα τόσο, ένα τόσο περίπλοκο θέμα με τόσο μεγάλη ικανότητα. Συμφωνώ λοιπόν με την ανάλυση την οποία κάνατε, αλλά ίσως να καταλήγω σε σχετικά διαφορετικά από συμπεράσματα. Έχω την αίσθηση ότι το σχέδιο οδηγίας το οποίο έχουμε μπροστά μας πρέπει να εξεταστεί στο σύνολό του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποτίθεται καλείται να παρουσιάσει ένα έγγραφο το επόμενο φθινόπωρο. Το έγγραφο αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποβεί επικίνδυνο. Είχα αρκετές συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτό και τίποτα δεν με έχει οδηγήσει μέχρι τώρα να αλλάξω τις θέσεις τις οποίες είχα καταλήξει από πριν. Υπάρχει ένα θέμα ανταγωνιστικότητας το οποίο τίθεται, όμως το επιχείρημα το οποίο ε, χρησιμοποιείται δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Θα μπορούσε να πει κανείς ε, και τι είναι οι συνέπειες, ποιες είναι οι συνέπειες για το περιβάλλον. Φαίνεται ότι οι συνέπειες για το περιβάλλον είναι σχετικά περιορισμένες, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να εμπλακούμε σε μία τόσο λίγα υποσχόμενη οδό για το μέλλον. Θα σας παρακαλούσα, λέει ο κύριος Κράμερ, να κοιτάμε την ώρα ε, πριν και μετά και να περιορίσουμε την ώρα ομιλίας ε, νωρίτερα, όχι να φτάσουμε στο παραπέντε που θα τελειώσουμε τώρα και να έχουμε τόσους ομιλητές. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι τηλεγραφικός πρέπει να προσέξουμε εδώ περί τίνος πρόκειται. Είναι ένα ελάχιστο ευέλικτο σύστημα για μία οδηγία κινητήρων μη οδικών. Απότερο στόχος μας είναι η ατμοσφαιρική ποιότητα. Τώρα σκέφτομαι αν πρέπει να γίνει αυτή η τροποποίηση ή όχι. Και το ερώτημα αυτό έχει τεθεί και από μία προηγούμενη συγγήτρια και από άλλους συναδέλφους. Νομίζω ότι όλη η υπόθεση αυτή της τροποποίηση της οδηγίας ξεκίνησε από διάφορα σιδηροδρομικά λόμπι, διότι υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την παρούσα οδηγία αλλά σε ορισμένα κράτη-μέλη θα πρέπει να σταματήσουν οι συνδρομικές μεταφορές εάν δεν δοθεί αυτό το μεγαλύτερο περιθώριο, αν δεν γίνει πιο ευέλικτο το σύστημα. Αυτό λοιπόν που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να υποχρεώσουμε τους μικρομεσαίους κατασκευαστές τέτοιων λοκομοτίβων ή κινητήρων να ε, υποκύψουν στις απαιτήσει ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους. Ή θα τα ε, περάσουμε αυτά για όλους ή για κανέναν. Και εδώ υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Αυτό το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε και είναι αυτό το οποίο προτείνει η συγγήτρια, είναι να επανακάμψουμε στις, στο, ευέλικτο στο ευέλικτο σύστημα του 2004. Μπορούμε να συζητήσουμε εάν διευρύνουμε το ευέλικτο σύστημα, ναι ή όχι, αλλά αυτό δεν μπορούμε να ξαναπροτείνουμε κάτι το οποίο ήδη υπάρχει στην νομοθεσία, δηλαδή τα συστήματα του 2004. Ο κύριος Φον Πάικεν. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Έχει, είναι τεράστιο το θέμα αυτό, έχει νομοθετικές α, ε, ε, επιπτώσεις και θα πρέπει τους νομοθετικούς φακέλους να τους έχουμε εγκαίρως στη διάθεσή μας και όχι τα τελευταία πέντε λεπτά ασχολείται με την ποιότητα του αέρα και όταν μιλάμε για την ποιότητα του αέρα πάρα πολλές ομάδες σε αυτό το κοινοβουλίο λένε ε, τα γνωστά, δηλαδή ότι απαιτούνται πολιτικές παρέμβαση στην πηγή. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε ακούσει και από τον Επίτροπο Ποτόσνικ να λέγει ότι δεν μπορεί να φτάσει ε, και να ελέγξει τα επίπεδα εκπομπών σε εθνικό επίπεδο αν δεν έχουμε σωστές πολιτικές επηρεασμού των πηγών. Τώρα λοιπόν συζητάμε τα θέματα των πηγών. Συζητάμε για κινητήρες ε, για μη οδική χρήση που αντιπροσωπεύουν το 7% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ε, και το 14% άλλων, άλλου τύπου ρήπαντων. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2004 ήδη είχαν αρχίσει οι συζητήσεις και χρειάστηκαν 7 χρόνια να ξεκινήσει η εφαρμογή. Και πάρα πολλές εταιρείες κινούνται ε, είναι αλήθεια ότι λένε ότι δεν είναι διαθέσιμες κάποιες ε, κάποιοι κινητήρες ε, για σιδηροδρομική χρήση δεν είναι αλήθεια αυτό. Στη Σουηδία ε, και στη Γερμανία είναι διαθέσιμες οι μηχανές αυτές και οι υπόλοιποι θεωρούν ότι φύγονται γιατί δεν έκαναν τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν δεν καταλαβαίνω ποια είναι η στάση μας. Μιλάμε εδώ για μια ουσιαστική πολιτική να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα και η επιλογή δεν είναι παρά μόνο ε, να απορρίψουμε ουσιαστικά τις προτάσεις οι οποίες δεν βοηθούν. το ο κύριος Κάλαχαν και μετά η κυρία Κλάς. Ευχαριστώ και εγώ λυπάμαι που δεν έχουμε επαρκή χρόνο να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό ντοσιέ, αλλά χαίρομαι που η Κομισιόν σημείωσε τις καταστροφικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και δέχεται να ε, τροποποιηθεί η οδηγία ε, για ε, να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του κινητήρες αυτούς. Θα χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που η Κομισιόν δέχεται να αλλάξει αυτό το ευέλικτο σύστημα και η αντιμετώπιση της είναι πολύ ρεαλιστική. Υπάρχει ένας μειωμένος αριθμός τέτοιων κινητήρων για τα οποία θα πρέπει να, πρέπει να ισχύει κάποια παρέκκληση και ε, δημιουργούνται ιδιαίτερες δυσκολίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που λαμβάνονται υπόψη αυτός ο αριθμός και οι τύποι κινητήρων, αν και θα ήθελα να καλυφθούν περισσότεροι τύποι κινητήρων σε αυτή την τροποποίηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί θέλει να εξαιρέσει τον οικοδομικό τομέα. Θα ήθελα και αυτός να περιληφθεί. Επίσης καταλαβαίνω ότι δεν θα πρέπει να υποβαρυνθούν, επιβαρυνθούν ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Ε, θα πρέπει να περιληφθούν και οι μεγάλες επιχειρήσεις στο ευέλικτο σύστημα. Η τροπολογία 10 ε, ε, αποκλεί του, τον οικοδομικό κατασκευαστικό τομέα από τις τροποποιήσεις αυτές ε, δεν συμφωνώ διότι πολλοί τέτοιοι κινητήρες χρησιμοποιούνται και στη δασοκομεία αλλά και στο, στην εξκαφή, στις εξκαφές, ε, μετακινήσεις ε, εδάφους ε, κλπ. Χρειαζόμαστε λοιπόν να συμφωνήσουμε γρήγορα για να περάσουν αυτές οι τροποποιήσεις των διατάξεων και γι' αυτό ε, βασίζουμε στις ε, επιτυχείς ενέργειες της εισηγήτριας. Ευχαριστώ η κυρία Κλάς. Ευχαριστώ. Ε, δεν είναι μεγάλο κλάδος αυτός, αλλά είναι σημαντικός. Δεν πρέπει να πάρουμε αποφάσεις συναισθηματικές αλλά ρεαλιστικές. Πράγματι, οι κατασκευαστές έχουν αρκετές δύσκολες με την προσαρμογή στο 3β. Πρέπει να κάνουν ορισμένες τεχνικές προσαρμογές. Από την άλλη, από τη μία πλευρά υπάρχουν τα ποσοστά των κινητήρων, από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι ε, κατασκευαστές των μηχανημάτων πρέπει να προσαρμοστούν όσον αφορά τις εκπομπές, ε, την ασφάλεια της εργασίας και της λειτουργίας και αυτοί οι κινητήρες ε, είναι, έχουν ιδιαιτερότητες. Γι' αυτό είναι σημαντική η ευελιξία, ένα ευέλικτο σύστημα, όχι μόνο για τις λοκομοτίβες, αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλος ο οικοδομικός κατασκευαστικός τομέας ε, χρησιμοποιεί αυτούς κινητήρες ε, και βασίζεται σε αυτούς και γι' αυτό ε, πιστεύω ότι αυτό το ευέλικτο σύστημα θα τους ωφελήσει ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Dziękuję pani Klas. Pani Katrin Suli, a następnym mówcą będzie pani Linda Makew. Κυρία Suli. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι προφανές η κρίση θίγει όλους τους τομείς, όχι μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μεγάλες επιχειρήσεις, την οικοδομή και η ανάκαμψη εκεί είναι πάρα πολύ χαμηλού επίπεδου. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω κυρίως την έλλειψη ευελιξίας που υπάρχει στους κινητήρες αντικατάστασης που θα επηρεάσει τις περιφερειακές, τα περιφερειακό δρομολόγια στην Γαλλία. Είναι μικρά δρομολόγια, μικρής διάρκειας και το κόστος ενημέρωσης των κινητήρων είτε μέσω τεχνικών αλλαγών είτε μέσω με την αγορά νέου υλικού θα επηρεάσει άμεσα τις τοπικές αρχές, στη συγκεκριμένη την περίπτωση της Γαλλίας οι περιφέρειες είναι υπεύθυνε και οι πολίτες οι οποίοι είναι χρήστες και επιβάτες φυσικά θα πληρώσουν το κόστος και πληρώνουν μάλιστα θα πληρώσουν δύο φορές το κόστος γιατί είναι και ε, χρήστες αλλά πληρώνουν και φόρο γύρω από αυτά. Το να αυξήσουμε λοιπόν τον φορολογικό βάρος των πολιτών μας δεν είναι κάτι το θετικό. Δεν θα πρέπει φυσικά να πούμε ότι θα αγοράσουμε υλικό το οποίο δεν θα είναι το απαιτούμενο επίπεδο, αλλά θα πρέπει να βρούμε μια κάποια άλλη λύση η οποία να επιτρέψει ε, στις ιοδρομικές εταιρείες να χρησιμοποιούν το παλαιό υλικό χωρίς ε, να προκαλέσουμε κόστη τα οποία δεν μπορούμε να καλύψουμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διερμηνείς που είναι στη διάθεσή μας ε, και μετά τις 6.30. Μακάβανε. Ε, το θέμα αυτό αφορά την, ε, ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι είναι διαθέσιμο σε επίπεδο μηχανών έλξης και κινητήρων μηχανών έλξης στους ιδιοδρόμους. Ξέρουμε ότι υπάρχουν εντελώς διαφορετικές συνθήκες στην Ευρώπη και υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά της Έχουμε αρχίσει να μην έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και δεν θα ακούσουμε προφανώς σήμερα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Ελπίζω να γίνει μια κάποια συζήτηση όταν θα έχουμε όλα τα δεδομένα στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Λίζε. Πρόεδρε, Σύμφωνα με αυτά που είπε η Λίντα Μακέβαν, ε, πρέπει να βρούμε χρόνο. Κάποτε είπαμε να συζητήσουμε και την έξεση του Σαλβατόρα Ταταρέλα. Ίσως λοιπόν θα μπορούσε η γραμματεία να βρει χρόνο και να το συζητήσει με τον πρόεδρο. Ε, τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα πρέπει να πω ότι το θέμα είναι τεχνικά δύσκολο. Έχω ακούσει διάφορες απόψεις, διάφορες εκδοχές. Κάποιος μάλιστα μου είπε ότι πριν από 8 χρόνια πίστευαν ότι αυτές οι τιμές δεν μπορούν ε, να, να εφαρμοστούν, δεν είναι εφαρμόσιμες. Βλέπω όμως τώρα ότι έχει ασκηθεί σωστή πίεση για να προχωρήσουμε περισσότερο και σε καινοτομίες. Αλλά κάτι πρέπει να παρατηρήσω. Η Κομισιόν έκανε ένα τεράστιο λάθος λέγοντας ότι σε ένα φάκελο ο οποίος εδώ ε, βρίσκεται στην αρμόδια επιτροπή επί της ουσίας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, πρωταρχικά την οικονομική κρίση. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να ξεπεραστεί η κρίση, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή τη βασική, ε, αυτό ως βασικό αίτιο. Ε, την οικονομική κρίση. Βασικά είναι το, η προστασία του περιβάλλοντος. Εκεί επικεντρωνόμαστε. Ευχαριστώ. Βεβαίως, μετά από αυτά που είπατε, θα τα θέσω αυτά υπόψη και ενδεχομένως να κάνουμε μια εκτακτή συνεδρίαση των συντονιστών. Η κυρία Κάντεμπαχ. Μιλήσαμε με τον Επίτροπο Ποτότσνικ για την ε, βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, νέες τεχνολογίες, οικονομική κρίση, επενδύσεις, καινοτομίες, τεχνολογία. Και μετά μιλάμε εδώ για την διεύρυνση της ευελιξίας λόγω της οικονομικής κρίσης. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αυτό βασικά με το στοιχείο του περιβάλλοντος και όχι με, την οικονομική, με στοιχείο της οικονομικής κρίσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρδίνη. Κυρία Γκαρδίνη, λίγες σκέψεις θα ήθελα να εκφράσω. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να εμβαθύνουμε στο θέμα είναι θέματα αρκετά περίπλοκα και τεχνικά και νομίζω ότι περαιτέρω ερεύνηση δεν θα αυλάψει. Το θέμα της κρίσης δεν είναι κάτι το αφηρημένο που αφορά την οικονομία γενικότερα, αλλά μιλάμε για αυξημένες συνέπειες στην αγορά εργασίας και θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Νομίζω ότι θα πρέπει λοιπόν να εμβαθύνουμε λίγο προς την κατεύθυνση αυτή γιατί υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιες προσπάθειες εδώ οι οποίες γίνονται, αλλά αναγνωρίζονται οι δυσκολίες που υπάρχουν σε τομείς όπως το σιροδρομικό υλικό, αλλά οι δυσκολίες αυτές δεν λαμβάνονται τελικά υπόψη. Εγώ νόμιζα ότι θα είχαμε περισσότερο χρόνο για να μπορέσουμε ε, για κάποιες κατηγορίες κινητήρων να καταλήξουμε νομίζω χωρίς πολλές συζητήσεις έτσι ώστε μετά από τρία χρόνια να περάσουμε στην φάση 4 από την 3β που βρισκόμαστε τώρα. Ίσως στο παρελθόν να έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη όταν καθορίστηκαν τέτοια περάσματα θα έλεγα σε διαφορετικού τύπου κύκλους παραγωγής για την απαραίτητη ευελιξία η οποία θα πρέπει να ισχύει για όλους. Νομίζω ότι μία θα έλεγα προσπάθεια καθορισμού του ποσοστού αυτού της ευελιξίας είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας προστατεύσει από ορισμένε καταχρήσεις γιατί υπάρχουν κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να καλύψουν ε, τα προβλήματα που υπάρχουν αλλά υπάρχουν όμως και ε, μικρότερες επιχειρήσεις που δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τις νέες ανάγκες και θα φυγούν οι μικρές επιχειρήσεις, θα λειτουργήσει το σύστημα υπέρ των μεγάλων. Πρέπει λοιπόν να είμαστε όλοι δίκαιοι και αποτελεσματικοί. E, termin składania poprawek 9 lutego do godziny 12, no biorąc pod uwagę sytuację, jaka się... E,